Αγαπητοί, μήπως θέλετε να καθίσετε για να επανακάμψουμε δρυμύτερες τις εργασίες μας. Θα ήθελα εξ ονόματός σας πρώτα απ' όλα να υποδεχθώ τον κύριο Χάινς Μπέκερ, εξ ονόματος όλων, ο οποίος είναι νέο μέλος της Επιτροπής μας από το ΕΛΚ και καταλαμβάνει ένα κενό εδόλιο Καλώς ήρθατε κύριε Μπέκερ. Είναι ένα μεγάλο προνόμιο αυτό γιατί δεν υπάρχει τόσο ενθουσιασμός όταν έχετε ένα νέο μέλος όπως στη δική σας περίπτωση. 17 σημείο της ημέρας διάταξης. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Στην θητεία μας με την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους σε σχέση με την οδηγία για το χρόνο εργασίας και την εφαρμογή της. Έχουμε ένα σημαντικό αριθμό προς και κλειμένων, αλλά επειδή κατανοώ ότι η Κομισιόν η οποία και αυτή εκπροσωπείται θα ήθελε να λάβει το λόγο και επειδή και ο εισηγητής μας που είναι ο εισηγητής της προηγούμενης θητείας. Ίσως θα ήθελε και αυτός να πει κάτι το εισαγωγικό. Όχι. Ε, εντάξει, μετά. Η Κομισιόν τότε. Ο κύριος Αρμίντου Σίλβα, ο οποίος είναι ε, ε ασκών την διεύθυνση σε κάποια υπηρεσία σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την ε, πρόσκληση στην Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και συμπερίληψη. Είναι πολύ καιρό που δεν έχει συζητηθεί το θέμα αυτό σε αυτή την Επιτροπή και γι' αυτό θα ήθελα απλώ να υπενθυμίσω ότι η οδηγία για το χρόνο εργασίας αποτελεί ο ακρογωνιαίο λίθο της ε, κοινωνικής Ευρώπης και έχει σαν στόχο να καθορίσει ανώτατα όρια για τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων σε εβδομαδιαίο και ημερήσιο επίπεδο, σε ετήσιο επίπεδο επίσης σε ό,τι αφορά την νυχτερινή εργασία και φυσικά υπόκειται και σε ένα μεγάλο βαθμό εξαιρέσεων και προνοιών ευελιξίας που μπορούν να γίνουν με νόμο με συλλογική σύμβαση ή σε περίπτωση αυτεξαίρεσης με την προσωπική συγκατάθεση του εργαζομένου. Αυτό ισχύει για όλους τους τομείς εκτός από αυτούς που καλύπτονται από ειδική νομοθεσία όπως είναι παραγωγικά ο τομέας των μεταφορών που καλύπτεται από ειδική νομοθεσία. Αλλά κατά άλλα έχει συνολική εμβέλεια. Μετά από την αποτυχία της συνδιαλλαγής το 2009 μεταξύ Συνοβουλίου και Κοινοβουλίου, η Κομισιόν ξεκίνησε αμέσως τη διαδικασία ε, αναθεώρησης οδηγίας 2003 88 με ένα τριπλό στόχο. Πρώτον, την προσαρμογή αυτής της νομοθεσίας για τον χρόνο εργασίας ε, στις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από νέα σχήματα εργασίας, νέες μορφές εργασίας, νέα σύνθεση της δύναμης εργασίας. Η παλιά οδηγία ήταν 20 ετής. Να μειωθεί επίσης η ανασφάλεια δικαίου ήταν η πρόθεση της Κομισιόν και να υπάρξει και μία πάγια νομολογία επειδή ορισμένε ρυθμίσεις είχαν τύχει αμφισβήτησης και επίσης να αντιμετωπίσει προβλήματα ολοσθήσεως σε ορισμένους τομείς και σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη διαδικασία αναθεώρησης με μια διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων το Μάρτιο του 2010 και ακολουθήθηκε αυτό από μια δεύτερη διαδικασία διαβούλευση το Δεκέμβριο του 2010 10, όπου ζητήσαμε και την άποψη των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με μια σειρά από συγκεκριμένε επιλογέ για τη μεταρρύθμιση τη οδηγία αυτή. Συγχρόνω, δημοσιεύσαμε εκτενή στοιχεία σε σχέση με τα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα αυτής της οδηγίας, την επίπτωσή της επίσης και επίσης σε σχέση με το στάδιο νομικής εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο αυτής της έκθεσης. Μία έκθεση λοιπόν εφαρμογής δημοσιεύσαμε και μια έκθεση που έγινε από ένα εξωτερικό σύμβουλο, την περιόνιμη εταιρεία Deloitte, την ίδια μέρα που η Κομισιόν ζήτησε την άποψη των κοινωνικών εταίρων. Είχαμε λοιπόν σαν στόχο να έχουμε πλήρη στοιχεία και στοιχεία ποιότητα σε σχέση με τις επιπτώσεις της οδηγίας. Η οδηγία, η έκθεση επιπτώσεως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλοί εργαζόμενοι στην Ευρώπη καλύπτονται από ελάχιστες προδιαγραφέ για τον χρόνο εργασία Σε ορισμένε χώρε οι προστατευτικέ που προέρχονται από συλλογικέ συμβάσεις ρυθμίσει, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά υπάρχουν συμβάσει, προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν και τα οποία καταγράφονται εξονυχιστικά στην έκθεση. Υπάρχουν ομάδες εργαζομένων που δεν καλύπτονται ακόμα επαρκώς έναντι υπερβολικών ορών εργασίας ή της υποχρέωσης να εργάζονται σε αντικοινωνικές, μη τυπικές χρονικές περιόδους. Επίσης είδαμε να υπάρχει έλλειψη εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομολογίας, ιδίως στα νοσοκομεία και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Είδαμε επίσης να υπάρχει πολυ, πολυπληθωρισμός στην αυτοεξαίρεση, η οποία ισχύει τώρα για 16 κράτη-μέλη, για 5 χώρες σε όλους τους οικονομικούς τομείς και σε άλλες 11 σε συγκεκριμένους τομείς για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει, προκύψει από την ε, νομολογία Σίμα Γέγκερ και επίσης έχουμε διαπιστώσει μια έλλειψη σαφήνεια στην εφαρμογή, στην ερμηνεία ορισμένων ασαφών στοιχείων στην οδηγία, όπως παραδείγματος το ότι είναι αυτόνομος εργαζόμενος, την εφαρμογή ε, σε περιπτώσεων πολλαπλών συμβολέων, ο συνδυασμός της άδεια με άδεια ασθένειες κτλ. Παρουσιάσαμε στους κοινωνικούς εταίρους δύο βασικές επιλογές σε σχέση με την αναθεώρηση. Είτε μια εστιασμένη αναθεώρηση που συγκεντρώνεται Συγκεντρώνω την προσοχή στα θέματα τα οποία παρά την ομολογία είναι ακόμα αδιαλεύκαντα, όπως είναι η καταμέτρηση του χρόνου εργασίας σε ατυπικές συνθήκες, ιδίως σε νοσοκομεία και σε πυροσβεστικές υπηρεσίες και επίσης το ερώτημα του ποια θα παίρνουν η χρονική στιγμή στην οποία δίδεται η αντισταθμιστική ανάπαυση. Όλα αυτά είναι σημεία στα οποία πρέπει να υπάρξει διασάφυνση των προνοιών που ισχύουν σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει τώρα φυσικά μια άλλη εναλλακτική προσέγγιση που είναι μια πλήρης συνολική μεταρρύθμιση η οποία πέραν αυτών των δύο θεμάτων προσπαθούσε να εξυγχρονίσει και να προσαρμόσει την τρέχουσα νομοθεσία. Δεν θέλω τώρα να είμαι εξαντλητικός σε αυτά που σας λέω, απλώς μπορώ να σας απαριθμίσω ορισμένα από τα θέματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει στην ανακοίνωσή μας. <clears throat> Είναι θέματα όπως η αυτοεξέρεξη, το opt-out δηλαδή, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιστασία των εργαζομένων που δέχονται να εργάζονται πάνω από 48 ώρες κατά μέσον όρο τη βδομάδα, το θέμα των αυτόνομων εργαζομένων, ο εξυγχρονισμός του ορισμού, ε, των ορισμών εν ώψη της ανάδυσης νέων μορφών εργασίας, το θέμα της ε, συμφιλίωσης οικογενειακής και εργασιακής ζωής, με τη δυνατότητα παραδείγματος χάρη να υπάρχει το δικαίωμα τροποποίηση του χρόνου εργασία από του εργαζομένου, επιπλέον η μεγαλύτερη ευκαμψία για την αντιμετώπιση νέων συνδικών εργασία και φυσικά και πάλι το θέμα του μήκους της περίοδου αναφοράς για να γίνεται μέσος όρος του χρόνου εργασίας, τι γίνεται στην περίπτωση των εργαζομένων που έχουν πολλαπλά συμβόλαια, αν θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνε σε κάθε συγκεκριμένη σύμβαση. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από προτάσει λοιπόν για τα θέματα αυτά και έχουμε υποβάλει την ανάλυση αυτή και την αξιολόγηση προς τους κοινωνικούς εταίρους. Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους τώρα περατώθηκε στις 25 Μαρτίου. Δεν έχουμε ακόμα μια πλήρη ανάλυση των περίπου 50 απαντήσεων που έχουμε λάβει από αυτή τη διαβούλευση. Το πιο σημαντικό σημείο το οποίο μπορώ να τονίσω εδώ για μένα είναι ότι η πιο σημαντική εγκάρση κατά κάποιο τρόπο κοινωνικοί εταίροι έχουν αναγνωρίσει την ειδική ευθύνη που επέχουν για να μπορέσει να εξευρεθεί μια λύση σε σχέση με την προσαρμογή της οδηγίας για, χρόνο, για το χρόνο εργασίας. Εκφράσανε τη θεληματικότητά τους να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις, αλλά χωρίς, προς το παρόν τουλάχιστον, να είναι σε θέση να συμφωνήσουν για το συγκεκριμένο πεδίο διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, εν γέννη, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν χαιρετήσει την δημοσίευση στοιχείων από την Κομισιόν σε σχέση με τα θέματα χρόνου εργασία και πολλοί από αυτού έχουν εκφράσει και την ικανοποίησή του με την ανάλυση η οποία προετάθη από την Κομισιόν παρά το γεγονό ότι μα επικρίνει και ορισμένοι από αυτού. Καταλήγουμε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου οι κοινωνικοί εταίροι αναμένονται να διαρευνήσουν και να βρουν κοινό έδαφος ώστε ή δυνατόν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, όταν είναι δυνατόν μάλλον. Εάν επιτύχουν συμφωνία λοιπόν για το πεδίο εφαρμογής, ελπίζουμε ότι θα το ε, διαβιβάσουν στην Κομισιόν με μία κοινή δήλωση και έτσι θα ξεκινήσει μια εννεάμινος περίοδος διαπραγματεύσεων. Εφόσον η κοινή υπάρξει μια συμφωνία στο τέλος αυτών των διαπραγματεύσεων από τους κοινωνικούς εταίρους, δίνανται και σίγουρα σε αυτήν την περίπτωση αναμένεται να το πράξουν, να θέσουν μια πρόταση στην Κομισιόν. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει αυτή τη συμφωνία για απόφαση του Συμβουλίου. Θα προκύψει μια οδηγία βάσει του άρθρου 155 της συνθήκης με πληροφόρηση του Κοινοβουλίου αλλά χωρίς μια επίσημη νομοθετική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν και αυτή είναι η προσέγγιση με την οποία η Κομισιόν έχει προβλέψει να γίνει η αναθεώρηση της οδηγίας αυτής για το χρόνο εργασίας. Ευχαριστούμε. Ξεκινάει η ακρόαση τώρα με τους κοινωνικούς εταίρους. Θα δώσω το λόγο σε αυτόν που μου προτάθηκε. Δηλαδή, η κυρία Ρεβέκα Σμιθ πρώτα, εκ μέρου του Business Europe. Μην ακολουθείτε πάντως το καλό και κακό παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιλήστε τόσο. 7 λεπτά. you, I'd like thank the... Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε και έτσι μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας και τις θέσεις μας. Στην Business Europe, όπως συμβαίνει και με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους στην Ευρώπη, βρισκόμαστε στη διαδικασία συζήτησης στο εσωτερικό μας του θέματος αυτού. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να σας πω ενδεικτικά πώς η Πρόεδρος διακόπτει. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε την ακρόαση αυτή στο γενικό της πλαίσιο. Βλέπετε, είμαστε στην αρχή της διαδικασίας, πράγματι. Ο συγητής πάντως και υπεύθυνοι των ομάδων σκέφτηκαν ότι ακριβώς γι' αυτό Τώρα που ξεκινάει η διαβούλευση για αυτή την υπόθεση, πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση με διαφάνεια, ώστε να συζητηθούν οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το πνεύμα σας καλούμε. Οπότε θέλουμε και περιμένουμε από σας να μας ε, μιλήσετε ακριβώς για τη συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό της οργάνωσής σας. Ακριβώς αυτό σκόπευα και εγώ να κάνω, λέει η κυρία Σμιθ, να σας παρουσιάσω πώς έχουν οι συζητήσεις σε εμάς σήμερα. Λοιπόν, περιεχόμενο τι πιστεύουμε για το περιεχόμενο της αναθεώρησης της οδηγίας. Ποιο θα πρέπει να είναι αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι η αναθεώρηση της οδηγίας πρέπει να περιοριστεί για να εξετάσει τα θέματα που τίθονται λόγω της νομολογίας που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσον αφορά ε, τι αιτήσει αποδοχέ. Στην διαδικασία αυτή έχουμε μπει, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δικιά μας εκτελεστική επιτροπή αποφάσισε να συστήσει τι πρέπει να διαπραγματευτούμε οι κοινωνικοί εταίροι. Γιατί είναι αυτή η προσέγγιση μας όσον αφορά το περιεχόμενο. Γιατί πιστεύουμε ότι τα θέματα ε, του χρόνου και της ε, άδεια ε, της αναρωτικής είναι θέματα τα οποία πολλές φορές μέχρι τώρα είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλαμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει εδώ και κάποια αντίφαση με ε, τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό πολλά κράτη-μέλη παραβιάζουν τελικά τις ρυθμίσεις. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι δεν πρόκειται μόνο για την υγεία στο δημόσιο τομέα, πρόκειται και για τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και η Business Europe θέλει να βρει μία λύση για την ε, περίπτωση αυτή, είτε πρόκειται για τον ιδιωτικό τομέα, είτε πρόκειται για τον δημόσιο. Επίσης, ε, για τις αιτήσεις άδειε. Και αυτό είναι θέμα το οποίο μέχρι τώρα έχει να κάνει με την εθνική νομοθεσία. Πάντως, η γνώμη μας είναι ότι η νομολογία ε, κοστίζει πολύ για να τεθεί σε εφαρμογή ο χρόνος ανάπαυσης, αν θεωρείται χρόνος εργασίας ή όχι. Πιστεύουμε ότι έτσι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο προσωπικό. Τα... Πρέπει επίσης να πληρώνετε ε, τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε άδεια την οποία δεν πήρε τελικά ο εργαζόμενος. Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις αξίζει να τονίσουμε ότι οι ρυθμίσεις, οι αποφάσεις του δικαστηρίου είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ήταν επιθυμητά. Και αυτό φαίνεται από την μελέτη αξιολόγησης. Πάντως, επικεντρωνόμενοι σε αυτά τα δύο θέματα, οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους. Γιατί αυτά είναι θέματα σημαντικά και για τους εργαζόμενους. Επίσης, όσον αφορά το περιεχόμενο, πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί το opt-out. Χρησιμοποιείται από 16 χώρες μέλη προς το παρόν και όπως είπε και στο δεύτερο στάδιο διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι ρεαλιστικό να ζητάμε στα κράτη-μέλη να μην χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή που έχουν. Είναι και αυτό ένα σημαντικό μέσο ευελιξίας που έχουν οι επιχειρήσεις για να μπορούν να καλύψουν τις διακοιμάνσεις και να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες έτσι όπως τις ζητούν οι πελάτες τους και να μπορούν να δουλεύουν και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί θέλουμε αυτή την ε, προσέγγιση, γιατί πιστεύουμε ότι οι επικεντρωνόμενοι σε αυτά τα δύο θέματα, δηλαδή την ανάπαυση και την πληρωμή της ετήσιας άδεια, αυτό είναι ένας ρεαλιστικός τρόπος για να προχωρήσουμε και να πετύχει η αναθεώρηση. Θέλουμε μια πραγματιστική, μια ρεαλιστική αναθεώρηση της οδηγίας. Δεν πιστεύουμε ότι αν υιοθετήσουμε μια ευρύτερη προσέγγιση θα έχουμε λύση. Και αυτό επειδή ακριβώς είναι διαφορετικές οι θέσεις των χωρών μελών, διαφορετικές οι απόψεις μεταξύ των ε, θεσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Ως κοινωνικοί εταίροι λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα εκείνα που μπορούμε πιο ρεαλιστικά να πετύχουμε ε, συμφωνία και πιστεύω ότι γι' αυτό πρέπει να περιοριστούμε στα δύο αυτά θέματα τα οποία σας ανάφερα. Συμπερασματικά, φυσικά και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία προέκυψαν στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης. Κατά τη γνώμη μας όμως δεν θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αναθεώρηση της οδηγίας. Πρέπει να μείνουν στις επιχειρήσεις και στους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο να προσπαθήσουν να βρουν λύση. Είναι σημαντικό να μην αγνούμε το γεγονός ότι πολλοί διακανονισμοί έχουν ισχύσει μέχρι τώρα και έχουν βοηθήσει να τεθεί καλά σε εφαρμογή οδηγία στους χώρους εργασίας. Πρέπει να αφήσουμε τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις να βρουν λύσεις win-to-win σε επίπεδο επιχείρησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους τους κοινωνικούς εταίρους νομίζω. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στα θέματα εκείνα τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να λυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι αυτά τα δύο που σα ανέφερα, ο χρόνο και, και η πληρωμή των αδειών. Ευχαριστούμε για την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Σωματείων η κυρία Βίπκε Ακμακ. Αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε στην ακρόαση για την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Μπορούμε παράλληλα να πούμε α, πάλι τα ίδια και δεν θα σας παραξενέψει αν σας πω ότι η θέση μας είναι πολύ συγκεκριμένη όσον αφορά την οδηγία αυτή για την τελευταία δεκαετία. Δεν έχουμε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με αιτήματά μας. Δεν θα σας παραξενεύσει αυτό. Τα σημεία δηλαδή που θα μου ακούσετε να τονίζω. Τονίζω καταρχήν ότι έχουμε μια οδηγία που βγαίνει από το χώρο υγείας και ασφάλειας και στηρίζεται σε διεθνείς προδιαγραφές. Στη δεύτερη διαβούλευση για τη γνωμοδότηση, επειδή η Κομισιόν δεν έλαβε υπόψη τα αιτήματά μας και δεν τήρησε και τις υποχρεώσεις της η Κομισιόν σε σχέση με τα πορίσματα της ε, αξιολόγησης επιπτώσεων. Ακούσαμε από την Κομισιόν ότι υπάρχουν δύο προτάσεις στο τραπέζι η επικεντρωμένη αναθεώρηση και μια πιο γενική αναθεώρηση. Εμείς θέλουμε μια πλήρη αναθεώρηση της οδηγίας. Αυτό που μας ανησυχεί πιο πολύ όσον αφορά τις προτάσεις της Κομισιόν, όπως φαντάζεστε, είναι να παραμείνει το opt-out, να επεκταθεί η περίοδος αναφοράς. Σχετικά με το opt-out καταρχήν. Η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της μας λέει ότι πολλές χώρες μέλη προσφεύγουν ήδη στο opt-out και έχουμε μια διάδοση του μέτρου αυτού. Η Κομισιόν θεωρεί λύση τη μείωση την ανάγκη χρήσης του opt-out. Στην αξιολόγηση επιπτώσεων ήταν σαφές ότι με επέκταση του χρόνου εργασίας αυξάνεται ο κίνδυνος για την υγεία του εργαζόμενου. Και όταν μιλάμε για προαιρετικά περισσότερο χρόνο εργασίας. Μια εβδομάδα των 40 ερών ή μια καλή εβδομάδα εργασίας να αφορά την υγεία και την ασφάλεια και την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ιδιωτική ζωής. Η θέση μας δεν άλλαξε ως προς το opt-out. Εμείς θέλουμε να σταματήσει αυτό το μέτρο. Περίοδοι αναφοράς τώρα. Η Κομισιόν επεκτείνει τις περιόδους στην ανακοίνωση αυτή λέει μπορεί να γίνεται περίοδο αναφράση και πάνω από 12 μήνε ανάλογα με τη Συμφωνία των Κοινωνικών και μέχρι 12 μήνε αν υπάρχει νομοθετημένη συμφωνία μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικού εταίρους. Αυτό δεν είναι επαρκής προστασία για τον εργαζόμενο. Όταν λέμε για περίοδο πάνω από 4 μήνε, αυτό πρέπει να περνάει μέσα από διαπραγματευμένη λύση. Και πρακτικά ξαναθέτουμε το ερώτημα, σε ποιους τομείς πραγματικά χρειαζόμαστε πιο μακρές περιόδους αναφοράς. Απάντηση ακόμα δεν πήραμε. Για τις εφημερίες. Η Κομισιόν λέει πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας. Όπως είπε και η νομολογία του Ευρωδικαστηρίου. Αλλά μετά ακούμε θέλουν, ότι θέλουν να υπολογίζουν διαφορετικά τις εφημερίες. Εμείς θεωρούμε ότι όλα είναι χρόνες εργασίας, ακόμα και η εφημερία. Έτσι πρέπει να υπολογίζεται. Και να συμφωνεί και με την απόφαση του δικαστηριού. Μερικές από τις προτάσεις της Κομισιόν είναι σωστές, αλλά επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση. Η αντισταθμιστική άδεια Φαίνομαι για το χρόνο αντισταθμιστικό για την ανάπαυση. Η αξιολόγηση επιπτώσεων μας λέει ότι η περίοδος ανάπαυσης δεν πρέπει να αναβάλλεται. Πρέπει η άδεια αυτή να λαμβάνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για μας αυτό είναι θεμελιώδες, να υπάρχει ισοδύναμη αντικατάσταση αυτού του χρόνου εργασίας. Δεν βλέπουμε διάσταση φύλου στις προτάσεις Πρέπει να υπάρχει ένα δικαίωμα για τον εργαζόμενο να μπορεί να ζητήσει αλλαγές στην κατανομή του χρόνου εργασίας τους. Βέβαια όλα αυτά τα έχει προωθήσει μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπολογίζουμε σε εσά να μας υποστηρίξετε σε όλα τα σημεία αυτά. Τώρα, τι πρότεινε η Κομισιόν στη δεύτερη διαβούλευση. Δεν βλέπουμε πραγματική αλλαγή πολιτικής τα χρόνια αυτά. Δεν βλέπουμε νέες προτάσεις. Συνεπώς αποφασίσαμε, και αυτό είναι το νέο στοιχείο όσο μας αφορά, οι διαπραγματεύσει των κοινωνικών εταίρων να ληφθούν υπόψη εφ' εξής. Εξού και το άνοιγμά μας για διαπραγματεύσεις αλλά με τους εξής στόχους. Θέλουμε μια πλήρη και συνολική αναθεώρηση της οδηγίας, να σταματήσει το opt-out στο εγγύς μέλλον, να έχουμε status quo στην αφορά της περίοδος αναφοράς και να υπάρχει συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου όσον αφορά τις, ταρεπό και τις εφημερίες. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η κυρία Λινιάν Πολίνσκι. Βολιζίνσκι. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας κυρία Πρόεδρε. Ναι. Ήρθαμε και πάλι εδώ σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που είναι ο χρόνος εργασίας. Και ξεκινάω λέγοντας ότι είναι μια σημαντική νομοθεσία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και για την ανάγκη για ελαστικότητα που ζητούν προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Θα περάσουμε στο περιεχόμενο των συζητήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προτείνονται διαπραγματεύσεις, γιατί είναι θέματα ζωτικής σημασίας για τους κοινωνικούς εταίρους. Και γι' αυτό και αποφασίσαμε και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Στην επόμενη μεταρρύθμιση της οδηγίας θα θέλαμε να αποφύγουμε να γίνει οδηγία πιο περίπλοκη από όσο ήδη είναι και από όσο ήδη είναι και οι εθνικές νομοθεσίες για το χρόνο εργασίας. Εμείς θέλουμε λύσεις που θα αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα βελτιωμένης ρύθμισης και που θα στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα αποφεύγει τη γραφειοκρατία και το περιττό άχθος για αυτές. Στην πρότασή μας για διαπραγματεύσεις Ξεκινήσαμε από τρία στοιχεία όσον αφορά το περιεχόμενο. Το πρώτο έχει να κάνει με την επίγουσα προτεραιότητα να ασχοληθούμε με τις περιπτώσεις που έχουν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τη νομική αβεβαιότητα που δημιουργείται. Εμείς αντίθετα θέλουμε βεβαιότητα για τις εφημερίες και για ε, την αντισταθμιστική ανάπαυση και για την πληρωμή της ετήσιας άδεια και της αναρωτικής. Θέματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχει εδώ ένα μπλέξιμο του τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό έχει να κάνει με την ελαστικότητα και το χρόνο αναφοράς. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι επίσης όρις όλες οι επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση ε, επιχειρήσεις που καλύπτονται από συλλογικέ συμβάσεις με άλλες μικρές επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από συλλογικέ συμβάσεις γιατί αυτές οι τελευταίες δεν έχουν περίοδο αναφοράς που θα ήταν οι 12 μήνες. Σήμερα, ιδιαίτερα μετά από την κρίση, να δούμε τη σημασία που έχει ο χρόνος ως ε, αναφορά για το χρόνο εργασίας το θέμα αυτό του, της αναφοράς, του χρόνου αναφοράς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύουμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η δυνατότητα χρήσης του opt-out, της ε, αυτοεξαίρεσης. Αν βέβαια έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη περίοδο αναφοράς, τότε αυτόματα θα περιοριστεί η χρήση της εξαίρεσης. Αυτό θα ήταν το σωστό. Γιατί λοιπόν ε, κάνουμε αυτή την επιλογή. Όπως είπε και η συνάδελφός μου από την Business Europe, αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε συμφωνία βάσει αυτών που μπορούμε να δεχτούμε γιατί έτσι θα υπάρχει μια ισορροπία και θα αποφύγουμε οποιοδήποτε παρατέρα μπλέξιμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τώρα Συνδικάτων Δημόσιας Δίκησης, ο κύριος ε, Ρίτσαρ Πού. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Η θέση μας αντικατοπτρίζει την θέση της ETUC, των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, οπότε δεν θα ήθελα να επαναλάβω, να επαναλάβω όλα αυτά τα πράγματα, απλώς θα επισημάνω ορισμένα επιμέρους σύμπια. Καταρχήν για το opt-out. Επαναλαμβάνω το προβληματισμό των σωματείων. Δεν θέλουμε να υπάρχει ε, η δυνατότητα αυτόνομης επιλογής της λύσης αυτής γιατί δεν υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού στην περίπτωση αυτή για όλη την Ευρώπη. Επίσης, ένα από τα μεγάλα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας είναι ότι οι δημόσιες αρχές και οι εργοδότες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την χρήση του opt-out για να έχουμε μια ρεαλιστική συζήτηση για την επέκταση του opt-out θα πρέπει να έχουμε νούμερα να συζητήσουμε. Νούμερα δεν έχουμε. Και αυτό είναι αποτυχία της εφαρμογής της νομοθεσίας. Η ανακοίνωση της Κομισιόν λέει ότι στο μέλλον θα υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση του opt-out. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με καλύτερη νομοθετική ρύθμιση και δεν είναι περίεργο που οι μικροί εργοδότες χαίρονται για το ότι δεν θα υπάρχει πιο στενή εποπτεία του συστήματος αυτού. Αν είχα μια ρεγιστική εικόνα του πώς και πόσο χρησιμοποιείται και σε ποιους τομείς και αν είναι ελεύθερο το άτομο να υπογράψει υπέρ αυτού ή όχι, αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο. Αυτά για το opt-out. Για τις εφημερίες, αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι υπάρχουν οι αποφάσεις του Ευρωδικαστηρίου και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποδυναμωθούν αυτές οι αποφάσεις και τα δικαιώματα. Πρέπει να έχουμε μια σύγχρονη προσέγγιση στο χρόνο εργασίας. Δεν έχουμε πιστεί για το ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στην οδηγία, διότι αν δούμε τις απαιτήσει σε 24 βάση στο δημόσιο τομέα. Πόσο δικημένεται ο χρόνος εργασίας στη γεωργία, στην βιοτεχνία, στη βιομηχανία. Όλα αυτά υπήρχαν πριν την οδηγία. Η οδηγία έχει την ευελιξία να καλύψει όλα τα επιμέρους αυτά σημεία. Δεν έχουμε πιστεί γιατί υπάρχει λόγος για αλλαγές. Όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, η νέα μέθοδος κυρίως στηρίζεται στην ισορροπία εργασία ιδιωτικού χρόνου. Αλλά η κρίση προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στον τομέα υγείας, είναι ότι τα άτομα εκεί δουλεύουν πολλές ώρες εφημερίες και περίεργες ώρες. Αυτά τα προβλήματα παραμένουν και τον επιμένουμε σε opt-out και σε αποδυνάμωση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε αντίθεση με την ιδέα ότι υπάρχει ανάγκη για μια σύγχρονη προσέγγιση στον χρόνο εργασίας. Έχουμε προγράμματα δράσης για προσλήψεις και λοιπά χρόνο εργασίας στα νοσοκομεία. είναι δυνατόν οι κοινωνικοί εταίροι στον κάθε τομέα να δουν επιμέρους τα θέματα αυτά και να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν. Την έκθεση Lloyds τώρα για τις ε, αξιολόγηση επιπτώσεων. Πρώτον, δεν έδωσε αποδείξεις υπέρ της θέσης της Κομισιόν και Υποστηρίζεται επιχειρήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ότι σε θέματα υγείας και ασφάλειας, ασφάλειας των ασθενών και ισορροπίας μεταξύ εργασίας και χρόνου ζωής έχουν δίκιο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αν δείτε το πώς διαδίδεται το opt-out, κυρίως είναι σε χώρες που χρησιμοποιείται στις δημόσιες υπηρεσίες και στην υγεία και αν μπορείτε να λύσετε το θέμα των εφημεριών με καινοτομίες όσον αφορά το opt-out δεν είναι μη ρεαλιστικό η χρήση του opt-out να είναι πολύ πιο περιορισμένη και μακροπρόθεσμα να καταργηθεί. Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων Γενικού κου ενδιαφέροντος και δημοσίου, ο κύριος Ανδρέας Πέρσον. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να σας μιλήσουμε. Θα σας περιγράψω τα κύρια σημεία για τις διαβουλεύσεις πρώτου και δεύτερου επίπεδου και τι γίνεται σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας η αγορά εργασία υπέστη σημαντικέ διαρθρωτικέ αλλαγέ τα τελευταία 20 χρόνια. Οι δημόσιε υπηρεσίε που δουλεύουν σε 24 βάση, η ανάγκη να παρέχονται αυτέ οι υπηρεσίε στο κοινό παραμένει. Οι προσδοκίε των πολιτών στο αφορά την ποιότητα και την ευελιξία των υπηρεσιών αυξάνεται. Οι δημόσιοι εργοδότε λοιπόν στηρίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό για να παρέχονται αυτέ οι υπηρεσίε. Αυτό ισχύει στον τομέα υγείας, στις, ε, στα επίγοντα περιστατικά κλπ. Και σε άλλους τομείς δηλαδή. Η γνώμη μας είναι ότι η μελλοντική αναθεώρηση του χρόνου εργασία χρειάζεται ισορροπία μεταξύ υγείας, ασφάλειας, ευελιξίας για εργοδότες και εργαζόμενους για καλή πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Βέβαια το θέμα των εφημεριών είναι σοβαρό πρόβλημα για το δημόσιο. Και όπω είπαμε στην απάντησή μα στη δεύτερη διαβούλευση, οι δημόσιε υπηρεσίε θα πρέπει να στηρίζονται στι ανάγκε του κοινού, να έχουν πρόσβαση στι ουσιώδει υπηρεσίε, πεσβεστική, υγεία, μεταφορέ, ε, υπηρεσίε ε, δημοσίου συμφέροντο σε 24 ώρε. Έπειτα χρειάζεται ισορροπία μεταξύ των αναγκών των χρηστών και τη ασφαλή και υγεία των εργαζομένων η οδηγία πρέπει να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των εργοδοτών του δημοσίου. Συμφωνούμε με το ότι δίνεται ιδιαίτερα έμφαση στις δημόσιες αρχές και στη φάση των διαβουλεύσεων από την Κομισιόν και στα συνοδευτικά έγγραφα. Τώρα η τρέχουσα διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας μετά από τη δεύτερη φάση διαβούλευσης για την αναθεώρηση Ήδη στην απάντησή μας στην πρώτη φάση είπαμε ότι υπάρχει δυνατότητα να πετύχουμε μια λύση με διαπραγμάτευση διατομεακά. Κατά τη γνώμη η οδηγία χρόνου εργασίας αφορά όλη την αγορά εργασίας και όχι επιμέρους τομείς μόνο. Τώρα το πεδίο διαπραγματεύσεων. Στην δεύτερη διαβούλευση στην απάντησή μας είπαμε ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των εφημεριών και τον ρεπό, αλλά και άλλα θέματα πρέπει να επιληθούν. Το πεδίο για τις διαπραγματεύσεις θα το αποφασίσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Εσωτερικά αυτή τη στιγμή συζητούμε τα επόμενα βήματα και κινήσεις μας. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον δικό μας εισηγητή αμέσως, χωρίς χρονοτριβή. Ευχαριστώ πολύ κύριος Θέρκας, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους μας για την παρουσίαση όλων αυτών των στοιχείων τα οποία μας διευκρινίζουν καλύτερα σε ποια φάση βρισκόμαστε και ποιες είναι οι ιδέες που πριτανεύουν σε αυτή τη δεύτερη φάση διαβουλεύσεων για μένα. Είναι το σημαντικό από τη δική μου πλευρά να σας ε, διαβεβαιώσω ότι το Κοινοβούλιο σέβεται πάρα πολύ τις διαδικασίες της ε, Συνθήκης της Λισαβόνας και γι' αυτό δεν πρόκειται να παρέμβουμε με κανένα τρόπο σε αυτή τη διαδικασία από προσωπική άποψη και κάτι που συμμερίζονται οι περισσότεροι συναδελφοί μου, νομίζω ότι είναι ότι αν υπήρχε κάποια στιγμή μια συνενετική λύση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων θα είχαμε καταφέρει να ξεπεράσουμε ένα ακαθόδες θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόμα. Για να γίνει όμω κάτι τέτοιο θα ήταν απαραίτητο οι, οι θέσεις οι οποίες ακούστηκαν σήμερα να διαφοροποιηθούν σε κάποιο βαθμό γιατί κάποιες απόψεις ήταν πραγματικά μαξιμαλιστικές άποψεις και βλέπουν μονάχα τη δική τους οπτική γωνία και εδώ χρειάζεται να δούμε πολυεδρικά το θέμα όλο των απόψεων για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ε, να μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε να υπενθυμίσω ότι η εμπειρία που συσσωρεύσαμε εδώ μας έχει καταδείξει ορισμένα σφάλματα τα οποία δεν πρέπει να επαναλάβουμε. Για μένα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό σε αυτήν την οδηγία να υπάρξει μια προσέγγιση των απόψεων για αυτή την οδηγία, γιατί βρισκόμαστε σε ένα περιοριστικό πλαίσιο, το οποίο είναι το πλαίσιο της ίδιας της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις, ε, τη διαδικασία νομοθετικών συμφωνιών μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού δίκαιο. Περιμένουμε ότι αυτή η οδηγία να επιτύχει ένα στόχο τον οποίο δεν ανέφερα ούτε η προσκεκλημένη μας ούτε η Κομισιόν. Ο στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτός είναι ο κυριότερος στόχος αυτής της οδηγίας. Θα υπάρξουν πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις, χάρη, για θέματα όπως είναι η πυρηνική ενέργεια. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε όταν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων πρέπει να το συζητήσουμε μέσα στα πλαίσια του θέματος της πυρηνικής ασφάλειας. Είναι χωριστό το θέμα του αν θέλουμε να έχουμε πυρηνική ενέργεια ή όχι. Ποιοι είναι οι κοινωνικοί στόχοι, τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις σε γενικές γραμμές. Όλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία είναι απόλυτα θεμητή. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι στενή η νομική βάση. Έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από την πρώτη στιγμή να θέτουμε στόχους οι οποίοι μπορεί να είναι συμπληρωματικοί ή δευτερεύοντες και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το βασικό θέμα που είναι η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. Ήθελα να πω επίσης στους προσκεκλημένους μας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζει πολύ καλά κάτι το οποίο προέρχεται και από την ίδια την ιστορία. Ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτα με το να παραγνωρίζουμε την ύπαρξη της Ευρώπης. Αυτό το θέμα έχει περάσει από δικαστήρια. Έχει γίνει κατηγορηματικά σαφές ότι η Ευρώπη έχει πραγματικά νομική υπόσταση και θα πρέπει να υπάρξει μια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ξεπερνάει τα εθνικά πλαίσια. Χρειάζεται να υπάρξει μια λύση για όλους τους Ευρωπαίους εργαζομένους οι οποίοι καλύπτουν τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν μπορεί ένα κράτος μέλος να έχει τα δικά του πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια που να υπολείπονται από αυτά τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επομένω, οποιαδήποτε προσπάθεια η οποία γίνεται να μην υπάρξει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ή το να υπάρχει μια εξαίρεση σε εθνικό επίπεδο <clears throat> ή να υπάρχουν επιμέρους εμβαλωματικές εξαιρέσεις δεν θα μπορέσει να επιτύχει. Ό,τι και να θέλουμε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει βάλει τον καθένα στη θέση του. Αυτό πρέπει να είναι σαφές σε όλους. Και τα κράτη τα οποία είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όταν τα κράτη μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουν ότι μπαίνουν σε μια κοινότητα αξιών. Ότι υπάρχει ένα κοινωνικό κεκτημένο. Ότι έχουν κάποιε υποχρεώσει σε σχέση με του ε, εργαζόμενου. Ότι υπάρχουν ελάχιστε προδιαγραφέ. Δεν είναι απλώ μια αγορά και μπάτε σκυλία, Λέστε, είναι μια ε, εν, οντότητα που έχει κοινοτικό χαρακτήρα και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Και για να κλείσω κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι όλοι οι βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλουν οι συνθήκες και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με τις διεθνείς συμβάσεις που έχουμε τόσο σεβασμό για αυτές για να μπορέσει σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχει μια ρύθμιση αυτών των θεμάτων θέλω να σας υπενθυμίσω γιατί και εγώ δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτά που ακούσαμε ότι δεν μπορούμε να διαφυσβητήσουμε την δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Το πρόβλημα είναι ότι η νομολογία του δικαστηρίου δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Πώς η Κομισιόν από το 2003 δεν έχει κάνει τίποτα για να επιτύχει την εφαρμογή αυτής της οδηγίας και δεν φέρνει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τα κράτη-μέλη τα οποία δεν τηρούν αυτή την οδηγία. Πώς υπάρχουν ε, εργαζόμενοι σε χώρες ορισμένες όπου δεν, ε, δεν τηρούν αυτά τα οποία αφορά η οδηγία. Γιατί δεν εφαρμόζεται η νομολογία αυτή, γιατί υποχρεώνται εργαζόμενοι να υπογράφουν συμβάσεις οι οποίες υπολείπονται από τι προδιαγραφέ τη Γιατί δεν έχει φέρει η Κομισιόν αυτά τα κράτη-μέλη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό είναι μια υποχρέωση που απορρέει από τι συνθήκε για την Κομισιόν. Τα κράτη λοιπόν-μέλη, τα οποία <clears throat> επανειλημμένα και κατά είναι έχουν παραβιάσει την οδηγία, θα πρέπει να βρίσκονται ενώπιον του Δικαστηρίου. Ακούσαμε τόσου υπεύθυνου, τόσου επιτρόπου να λένε ότι διαπραγματεύονται, ότι συζητούν με τα κράτη-μέλη, Άλλες φορές περιμένανε να γίνει μια τελευταία διαπραγμάτευση extremis και να υπάρξει μια συνενετική λύση. Αυτά τα ακούμε βερεσέ από το 2003. Οχτώ χρόνια. Οχτώ χρόνια είναι αυτά. Και δεν τηρείται η κοινοτική νομοθεσία. Κανείς δεν πράττει αυτά τα οποία είναι υποχρέωσή του να κάνει για να τηρηθεί η κοινοτική νομοθεσία. Η ενωτική, ενωσιακή νομοθεσία. Τέλος κυρία Πρόεδρε. θα ήθελα να δώσω μια πιο αισιόδοξη νότα. Ίσως μερικές φορές η ευφυΐα μας οδηγεί στο να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά πρέπει πάντα να τρέχουμε και κάποια αισιοδοξία. Εγώ άκουσα με μεγάλη με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπαν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα πλαίσιο για να υπάρξουν λογικές λύσεις σε όλες αυτές τις διαμάχες. Για πρώτη φορά άκουσα να μιλάνε για την ανάγκη των επιχειρήσεων αυτών να έχουν ευελιξία και για τους πολλαπλούς δρόμους που μπορούν να οδηγήσουν στην ευελιξία. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει σαφές και για το σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της αγοράς. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν μονάχα με μια ιδεολογική αντιμετώπιση. Πρέπει να υπάρχει ένα μέγιστο όριο στο χρόνο εργασίας στην Ευρώπη για κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να έχουμε όμως ευελιξία σε αυτά τα πράγματα. Το κοινοβούλιο, μπορούμε να έχουμε ευελιξία μάλλον στο θέμα αυτό, το κοινοβούλιο προέτεινε λύσεις οι οποίες ήταν ευέλικτες και μπορούμε να επαναλάβουμε αυτές τις προτάσεις μας. Και θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να ξεχάσετε τις μαξιμαλιστικές αντιμετωπίσεις για να λυθούν και τα προβλήματα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που συνδέονται πολλές φορές με την υπερβολική ε, ευελιξία. Το θέμα τώρα των εφημεριών. Μπορεί να υπάρξει μια επίλυση του προβλήματος που υπάρχει σε ορισμένε μορφές εργασίας, η συμφόρηση η οποία, η οποία προέρχεται από το θέμα αυτό των εφημεριών, αν εφαρμοστεί η απόφαση του δικαστηρίου. Μπορούμε όμως να βρούμε τη δυνατότητα λύσεων στα θέματα αυτά. Υπάρχουν αυτά τις οδηγίες που επιτρέπουν σε ορισμένες περιπτώσεις οι οικοί τομείς να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά με ad hoc λύσεις. Αλλά δεν πρέπει να ζητήσετε να γενικευτούν αυτές οι λύσεις. Ο στόχος μας είναι να λύσουμε προβλήματα, όχι να δημιουργήσουμε περαιτέρω προβλήματα. Και θα ήθελα να σταματήσω εδώ πρωτού με διακόψει η πρόεδρος. Θα ήταν ανώφελο να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα γυρίζοντας πίσω στο χρόνο την εποχή που δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν υπήρχε χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων ή να γυρίσουμε ένα αιώνα πίσω στο παρελθόν ή δύο, δύο αιώνες πριν όταν δεν υπήρχαν συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων και συλλογικές συμβάσεις. Λοιπόν, όταν δεν υπήρχαν κανόνες και όταν δεν υπήρχαν ε, ενώσεις εργαζομένων Αυτά τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν αυτές οι δομές και δεν πρέπει να ακολουθήσουμε ένα τέτοιο δρόμο προς το παρελθόν, πρέπει να βρούμε έναν δρόμο προς το μέλλον. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Σίγτα. Θα έλεγα, αυτοί που θα πάρουν το λόγο μετά από εσά να μην μακρηγορήσουν όπως και κάποιοι από τους προλαλήσαντες. Η κυρία Σρέτερ πρώτα. Παρακαλώ. Και εγώ πρέπει να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι καταλαβαίνω τη συγκινησιακή αντίδραση του εισηγητή. Αυτό το οποίο μας είπε η Κομισιόν είναι προκλητικού χαρακτήρα. Από τα πιο προκλητικά πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει σε αυτό το κοινοβούλιο και εγώ μπορώ να καταλάβω πολύ καλά γιατί αντιδρά με τόση αγανάκτηση ο κύριος ε, Θέρκας. Η Κομισιόν στην παρέμβασή της δεν είπε λέξη για την ασφάλεια της, ε, στην εργασία και την υγεία στην εργασία. Ούτε μία φορά η Κομισιόν δεν αναφέρθηκε στο ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το γεγονός ότι το Κοινοβουλίο είχε σταθμίσει μια κοινή θέση η οποία δεν έγινε δεκτή στη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά το Κοινοβούλιο είχε μια θέση. Και επίσης δεν ανέφερε το θέμα της νομικής βάσης που έχει να κάνει με αυτή την, ε, με αυτή την οδηγία. Σε αυτά τα οποία υπέβαλε γραπτός η Κομισιόν, δημιουργήθηκε σε μένα η εντύπωση ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι αν, αν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι ε, περνάνε στο σταυροδρόμι με κόκκινο, τότε η καλύτερη λύση είναι να, να να ρίξουμε το φανάρι, να το βγάλουμε από τη μέση και ας κόψουν το λαιμό τους οι πεζοί οι οποίοι πρέπει να περάσουν και αυτοί το δρόμο. Δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι λύση αυτή το να αφήσουμε τους εργαζόμενους χωρίς καμία προστασία της υγείας και της ασφάλειας τους. Αναφέρθηκε το θέμα των νοσοκομείων και των ε, πυροσβεστών, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και ασφάλειας. Χρειαζόμαστε μια, ένα πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίσει μια ουσιαστική προστασίας υγεία των εργαζομένων και δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα με την αυτοεξαίρεση, με τα opt-out. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε ουσιαστικά τον πυρήνα αυτής της νομοθεσία. Υπάρχουν κράτη τα οποία αυτή τη στιγμή αμφισβητούν τον χαρακτήρα της ίδιας αυτής της οδηγίας που έχει σαν στόχο την προστασία της υγείας και τις ε, ασφάλειες. Ενώ εμείς αυτό το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε είναι να καταλάβουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτά τα οποία λέει η οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια μέσα στις τωρινές συνθήκες. Αλλά είναι το α και το ω. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων έχουμε πάρα πολλές ε, μελέτες που καταδεικνύουν ότι όταν κάποιος ε, πρέπει να εργάζεται περισσότερες ώρες αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση που θέτει την υγεία του σε κίνδυνο με πολλαπλούς τρόπους. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη στην Ευρώπη με την μεγάλη αυτή οικονομία της Ευρώπης να βρούμε μια λύση και να δούμε με ποιους τρόπους θα έχουμε λύσεις έστω και ενδιάμεσες γιατί το ότι διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση σημαίνει αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος και μετά ο κύριος Τόμας Μάν. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα έλεγα ότι έχω γίνει τώρα πιο αισιόδοξο έχοντας ακούσει τους ε, κοινωνικούς εταίρους και τους συναδέρφους, κάθε άλλον. Μάλλον πιο σκεπτικιστής έχω γίνει από ό,τι κατά το παρελθόν. Έχοντας ακούσει ποια είναι τα διάφορα συμφέροντα που βρίσκονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους και οι διάφορες αξίες, είναι πράγματα που τα έχω ακούσει ξανά και ξανά. Δεν άκουσα τίποτα καινούριο. Δεν βλέπω γιατί γίνεται αυτή η προσπάθεια, γιατί περιμένουμε ότι θα πετύχει περισσότερο από ό,τι οι παλιότερες προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μόνο που βλέπω είναι ότι θέλουμε να κάνουμε διάφορες δηλώσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, θεαματικές και τίποτα παραπάνω. Η εκπρόσωπος της Business Europe, μάλιστα, θα λέγω ότι ήταν πιο επικοδομητική γιατί είπε ότι πρέπει αν μη τι άλλο να εντοπίσουμε τα σημεία πάνω στα οποία μπορεί να επιτευχθεί κάποια πρόοδος και πρέπει να επικεντρωθούμε στα σημεία εκείνα όπου μπορεί να γίνει ένα βήμα προς τα μπρος. Αν ε, το πετύχουμε αυτό, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Μια λοιπόν που συζητάμε αυτά τα θέματα, ας τα συζητήσουμε με κάθε λεπτομέρεια. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα σε αντιπαράθεση. Όπως υπάρχει από τη μια μεριά η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, και από την άλλη μεριά υπάρχουν ε, οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στα κράτη-μέλη. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χρειαζόμαστε ρυθμίσεις περισσότερο σε βάθος, με περισσότερες λεπτομέρειες για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως είναι η ε, ανεξάρτητοι αυτόνομοι επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή ψεύτο ελεύθεροι επαγγελματίες, να ξέρουμε για τις άδειε, τις αιτήσει, τις αναρωτικές. Υπάρχουν δηλαδή όροι που χρησιμοποιούμε για τους οποίους δεν έχουμε συγκεκριμένους ορισμούς, για να μην πω ότι μερικές φορές οι ορισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιφατικοί μεταξύ τους. Είναι λοιπόν ένα πακέτο για το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε συγκριτικές μελέτες. Θα έπρεπε να βαθύνουμε περισσότερο σε βάθος, να μάθουμε καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα, τότε μπορούμε να φέρουμε καλά σε πέρα στις, ε, την αποστολή μας. Το θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών δεν μας δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί μερικές φορές είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν σαν μισθωτοί, αλλά επίσημα τυπικά είναι εκείνοι υπεύθυνοι σαν να είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες, ενώ ακολουθούν τις οδηγίες κάποιου άλλου. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να δώσουμε σαφείς προσανατολισμούς στην ε, ρύθμισή μας. Αυτό πρέπει να το λύσουμε. Πρέπει επίσης να λύσουμε και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε τον χρόνο εφημεριών. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Βέβαια μερικές φορές ορισμένοι προτιμάνε να το αποφύγουν, να μην το λύσουν. Κάτι άλλο για το οποίο ούτε εδώ βλέπω τίποτα καινούριο είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια φορά μιλάει για την ευελιξία και ασφάλεια. Μιλάει για μια πιο ελαστική αγορά εργασίας. Έχουμε κάνει συζήτηση στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2020 και είπαμε ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, άρα πιο ελαστικοί στην εργασία, χωρίς όμως να έχουμε πει τι ακριβώς εννοούμε με αυτό. Και δεν είναι σύμπτωση αν 16 χώρες ε, χρησιμοποιούν το opt-out, την αυτοεξαίρεση, και άλλες χώρες μέλη χρησιμοποιούν άλλους δρόμους, είναι δημιουργικοί και βρίσκουν άλλες διεξόδους. Εγώ νομίζω ότι έχουν βρεθεί πολλοί τρόποι διαθέτησης του χρόνου εργασίας σε διάφορες χώρες, με ιδιαίτερη ελαστικότητα. Εδώ πρόκειται για συναπόφαση. Συνεπώς, πρέπει να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Αν, επαναλαμβάνω, 16 χώρες υιοθετούν μία θέση η οποία διαφοροποιείται από τη δικιά μας, ε, δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Έχουμε υποχωρήσει, έχουμε κάνει πολλές υποχωρήσεις. Πετύχαμε κάποιους συμβιβασμούς δύσκολους που μας πονάνε όλους. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κι άλλες υποχωρήσεις. Εξάλλου δεν υπάρχει κάτι που να μας ενθαρρύνει σήμερα από αυτά που ακούσαμε, οπότε ειλικρινά δεν βλέπω πώς μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Τέλος, πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη, να ενθαρρύνουμε και τους αυτούς μας, προκειμένου να δώσουμε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τους τομείς εκείνους που δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί. Εκεί δηλαδή όπου χρειαζόμαστε πιο ξεκάθαρες ιδέες για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Πρέπει να εντοπίσουμε δηλαδή πράγματι τους τομείς εκείνους στους οποίους υπάρχει ακόμα κάποια ευκαιρία να επιτευχθεί συμφωνία. Είναι περιτό να πετάμε άλλο ένα πυροτέχνημα το οποίο θα καταλήξει σε μια θεαματική αποτυχία εφόσον δεν υπάρχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να πετύχουμε αποτελέσματα. Δεν χρειάζονται διαβουλεύσεις αν δεν είμαστε πιο δημιουργικοί. Ναι στις διαβουλεύσεις αν είμαστε όμως αποφασισμένοι να πετύχουμε στην πράξη αποτελέσματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ωραία. Ο κύριος Τόμας μετά και ο Σκάρτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Βέρνερ από την ΕΤΟ είπε ότι είναι σαν να έχουμε, ξαναβλέπουμε το ίδιο έργο, σαν ένα déjà vu. Και πολλοί συνάδελφοι είπαν το ίδιο, ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Όπως είπε και ο κύριος Σάμπα, τα ίδια πράγματα βλέπουμε τα τελευταία 8 χρόνια με επαναλήψεις τελετουργικού χαρακτήρα. Αλλά φυσικά αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι σε πολλά κράτη-μέλη είχαμε διαφορετικές εμπειρίες και δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Αλλά το πλαίσιο πρέπει να παραμείνει ως πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Δεν είναι εύκολο. Θέλουμε, είπαμε, να υπάρξει μια συνολική επανεπεξεργασία της ε, οδηγίας αυτής δεν μπορεί να παραμείνει το business as usual και οι κανονισμοί για το opt-out, την αυτοεξαίρεση, φυσικά θα πρέπει να παραμείνουν γιατί αυτή τη στιγμή 16 χώρες αυτή τη στιγμή έχουν μια αυτοεξαίρεση και αυτό ισχύει μέχρι να υπάρξει κάποια διαδικασία επί παραβάσεως ε, και ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο το οποίο θα ακυρώσει αυτές τις αυτοεξαιρέσεις. Λοιπόν, στην πράξη πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Είχαμε και στο παρελθόν μια διαδικασία συνδιαλλαγής. Προσπαθήσαμε να βρούμε σημεία επαφής σε αυτή τη διαδικασία. Ίσως μια ισχυρή γέφυρα να φαίνεται ότι είναι ισχυρή, όπως αυτή η γέφυρα του Golden Gate στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά στην Ιαπωνία είδαμε τι μπορεί να κάνει ένα τσουνάμι. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι σταθερό. Προσπαθήσαμε παρόλα αυτά να έχουμε μία λύση για τα θέματα αυτά και εγώ ελπίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ευκαιρία για λύση. Κύριε Βέρκεν, είπατε ότι θα θέλετε να έχετε μία συγκεκριμένη ατζέντα τι γίνεται με τους νοσοκόμους, με τις νοσοκόμες, οι οδηγοί των ασθενοφόρων που δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες. Λοιπόν, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι βοηθοί νοσοκόμου. Λοιπόν, μπορείτε να εξασφαλίσετε την ισότητα των φύλων σε όλα αυτά τα επαγγέλματα, μπορούμε σε όλες τις ειδικότητες να εξασφαλίσουμε ισότητα των φύλων. Ένα δεύτερο ερώτημα στον κύριο Σίλβα από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις. Το καταλαβαίνω. Αλλά βλέπω και πάλι ότι σε πολλές διαβουλεύσεις, σε πολλές διαδικασίες αυτές που έχουν γίνει, στο τέλος όλα αυτά τα οποία έχουν βγει από τις διαβουλεύσεις ουσιαστικά δεν τα λαμβάνετε υπόψη στη συνέχεια. Γίνεται μια προσπάθεια να τα συνδέσετε όλα αυτά τα οποία βγάζετε από τις διαβουλεύσεις. Πώς προσπαθείτε να τα συνδέσετε με τη διαδικασία, πόσο στα σοβαρά παίρνετε αυτές τις διαβουλεύσεις. Αυτό είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε και λόγω της πίεσης χρόνου θέλω να ε, κλείσω με το εξή. Ο κύριος ε, Θέρκας αναφέρθηκε με το θέμα, στο θέμα των εφημεριών. Είπε ότι υπάρχει δυνατότητα να επιληθεί το θέμα αυτό και όχι με μια αυτοεξαίρεση που να βγαίνουμε τελείως από το πλαίσιο της οδηγίας. Είπε ότι υπάρχει μια λύση αν μπορέσουμε να είμαστε εύκαμπτοι κατά τομής. Είναι αυτό λοιπόν μια δυνατότητα που μπορούμε να την εφαρμόσουμε και σε άλλους τομείς, ώστε να υπάρξει μια ειδική λύση σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένους τομείς, διατηρώντας πάντα το γενικό πλαίσιο, δηλαδή να υπάρξει μια ευελιξία η οποία όμως μπορεί να γίνει πραγματικότητα εάν συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι για κάτι τέτοιο. Μήπως αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ε, οδό διαφυγής από το αδίέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε και θα θέλαμε να υπάρξει και ένα βήμα προς το εμπρός, να συνεχίσει ο διάλογος για τα θέματα αυτά και ίσως, όπως είπε και ο κύριος Θέρκας, να βρούμε έναν τρόπο να επιτύχουμε περισσότερη ευκαμψία χωρίς να καταστρέψουμε το συνολικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλάρ και η κυρία Γραμμιδαλή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούμε ευχαρίστηση ότι η έκθεση της Κομισιόν μας λέει ότι 16 χώρες από τις 27 εξακολουθούν να προτιμούν το opt-out. Αυτό είναι μια πλειοψηφία που μπλοκάρει και μερικοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτό στο παρελθόν. Κάποιος άλλος ομιλητής είπε ότι θα πρέπει να παραμείνει το opt-out. Συμφωνώ, αν 16 χώρες το θέλουν, θα πρέπει. Αυτό κάτι λέει για το opt-out. Οι χώρες έχουν επεξεργαστεί δική τους θέση ώστε να την απασχόληση και θα πρέπει να εξακολουθήσει αυτή η παράδοση να ισχύει. Το δεύτερο σημείο είναι οι εφημερίες. Έχει ιδιαίτερη επίπτωση στο ιατρικό επάγγελμα. Δεν ξέρω για τις εφημερίες, για τους οδηγούς φορτηγών κλπ. Ξέρουμε τι ισχύει εκεί. Ξέρετε όμως ότι στον Ηνωμένο Βασίλειο, και δεν μιλάω για άλλη χώρα, πέρυσι εκατοντάδες γιατροί έφυγαν, εγκατέλειψαν το επάγγελμα, γιατί πήγαν στα νοσοκομεία να κάνουν κλινική εκπαίδευση. Αλλά η οδηγία τους υποχρεώνει να αφήσουν αυτές τις κλινικές ώρες εργασίας πριν έχουν την αναγκαία εμπειρία και δεν μπόρεσαν να κάνουν την ειδίκευσή τους. Αυτοί οι δικαιωμένοι γιατροί δεν είναι όσοι πειραμένοι γιατροί με τους οποίους δούλευαν που κάνουν την κύρια δουλειά. Μάθαιναν, άκουχαν, βοηθούσαν. Πώς είναι δυνατόν να πούμε ότι η επέκταση των νερών θα αποτελεί πρόβλημα υγείας για αυτούς και περισσότερο πρόβλημα υγείας για τους ασθενείς. Χάσαμε εκατοντάδες πολύ νέους καλούς γιατρούς γιατί δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τη μία μέρα την άλλη. Γι' αυτό δεν είναι καλό για την υγεία και την ασφάλεια του πληθυσμού γενικότερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκριμαντέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τις ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να έχουμε εξαιρέσει. Σε ποιο κόσμο θέλουμε να ζούμε. Να δουλεύουμε περισσότερο, να κερδίζουμε λιγότερα και επιπλέον να να επιδεινώσουμε την υγεία μας στην εργασία, σε τι κόσμο θέλουμε να ζούμε. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, συμφωνώ με τον κύριο Θέρκας, χρειάζεται ένα μίνιμουμ σεβασμού της οδηγίας. Η μη τήρηση της οδηγίας, σε αντίθεση με αυτά που είπε ο προηγούμενος συνάδελφος, έχουμε 15 χώρες που δεν τηρούν αυτή την οδηγία είναι ξεκομμένες από την πραγματικότητα οι χώρες αυτές. Έπειτα έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο έχει πάρει ήδη απόφαση. Σήμερα για μένα είναι σαφές και αναγκαίο, το είπε ο κύριος Σέρκας, η υγεία και η ασφάλεια πρέπει να είναι στο κέντρο αυτής της οδηγίας. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ο κύριος Στίβεν Χιούτζ και μετά ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι κοινωνικοί εταίροι μακάρι να έχουν επιτυχία. Αν και το πρώτο εμπόδιο είναι η διαπραγμάτευση του πεδίου των διαπραγματεύσεων. Το πρώτο εμπόδιο. Και τότε χρειάζεται ευελιξία αν δούμε την οδηγία, ήδη υπάρχουν εξαιρέσεις κατά τομείς και κατά επαγγέλματα στην οδηγία. Στις ε, δεκαετία των 90 των η οδηγία, ήμουν ήδη ευρωβουλευτής. Τα κράτη μέγιστη διαπραγματεύσει τότε θέλανε η οδηγία να είναι πολύ ευέλικτη. Γι' αυτό έχουμε τις περιόδους αναφοράς, Γι' αυτό έχουμε τις εξαιρέσεις, το αρχικό άρθρο 17. Στο τελευταίο πακέτο προτάσεων προς το Συμβούλιο, όπως είπε ο Τόμας Μαν, προτείναμε επέκταση της περίοδου αναφοράς και επικρίναμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αλλά δεν ήταν επαρκές αυτό, διότι η χώρα μου και άλλες χώρες δεν θέλουν κανένα καθεστώς που να διέπει το χρόνο εργασίας θέλουν την άκρα ευελιξία. Κανέναν έλεγχο του χρόνου εργασία. Και αυτό ισχύει για εκατομμύρια Βρετανούς εργαζόμενους. Το δέχονται αυτό υπογράφοντα το συμφώνιο εργασία του και επεκτείνει και στι άλλε χώρε δυστυχώ αυτό. Και έχουμε στο βασικό σημείο κάτι που είπε η Ελίζαμπεθ με την ερώτησή τη. Η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακα των συνθηκών από το 2003, όπως είπε ο Τόμας και άλλοι. Είναι αλήθεια ότι το μόνο βήμα της Κομισιόν είναι διαδικασία παράβασης κατά κρατών μελών και θα ήθελα ο κύριος να μας πει τι γίνεται, τι κάνει η Κομισιόν σε σχέση με διαδικασίες παράβασης ως προς τις χώρες μένες που παραβαίνουν την οδηγία. Στο Βρετανικό δίκαιο υπάρχει ένας όρο που το λέμε judicial review, δηλαδή ένας φορέας μπορεί να ζητήσει από τα δικαστήρια να αποφανθεί κατά πόσον υπήρξε παράβαση του νόμου. Δεν ισχύει αυτό στην Ευρώπη, όπου η Κομισιόν μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το κατά πόσον υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ ενός μόνιμου opt-out για προστασία σε σχέση με την νομοθεσία υγείας και ασφάλειας έρχονται άνθρωποι εδώ μέσα και μας ακούνε και θα παραξενεύονται. Μιλάμε για νομοθεσία υγείας και ασφάλεια και λέμε 16 χώρε ζητανε ζητάνε opt-out από εξαίρεση. Αυτό είναι τελείω παράλογο. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να μπορεί η Κομισιόν να ελέγξει αυτή την ασυμβατότητα, να ζητήσει να ελεγχθεί από ένα δικαστή. Ο κύριο Κρίστενσεν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τους κοινωνικούς εταίρους για τις παρουσιάσεις τους. Φοβούμαι όμως ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αδιεξόδου. Αυτό φαίνεται και από τις διάφορες παρεμβάσεις. Είναι παράδοξο, αν μη τι άλλο, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι χώρες που δεν τηρούν τους ε, κανόνες, τις προδιαγραφές, τις οδηγίες, πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Ενώ δεν υποστηρίζουμε τα άτομα εκείνα τα οποία αγωνίζονται για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας. Οπότε, εσείς οι κοινωνικοί εταίροι, αν εσείς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμείτε να βρεθούν λύσεις για το χρόνο εργασίας, για την ασθένεια, για ε, τις εφημερίες. Αν θέλετε, πείτε μου, είναι λογικό να δουλεύει κανείς πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα, μάλιστα όλο το χρόνο. Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς που δικαιολογούν κάτι τέτοιο, που το αιτιολογούν. Η κυρία Λεκεβιτσέτη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήταν πολύ σημαντικό που βάλαμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας και θα θέλαμε να διαπιστώσουμε πρόοδο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Ακούσαμε τις απόψεις σήμερα των κοινωνικών εταίρων, τους ευχαριστούμε που ήρθαν. Ακούμε βέβαια διστάμενες απόψεις. Κάποιοι κοινωνικοί εταίροι υποστηρίζουν τις θέσεις Α, κάποιοι άλλοι τις θέσεις Β. Άρα είναι δύσκολα τα πράγματα και θα δυσκολευτούμε πολύ να καταλήξουμε σε συμβιβαστική θέση. Όλοι όσοι εργάζονται στις 27 χώρες θέλουν κάποια λύση. Εμείς όταν το 2004 η Λιθουανία δηλαδή μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ μάλιστα ήμουν τότε υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας και είχα την δυνατότητα να συνεργαστώ πολύ με τους κοινωνικούς εταίρους στη Λιθουανία. Και κάθε φορά αναγκαζόμασταν να ψάξουμε και να βρούμε συμβιβασμούς. Δεν μπορεί να λες ότι πρέπει να γίνονται υπερορίες στην Ευρώπη και τις υπερορίες πρέπει να την κάνει ένας εργαζόμενος ο οποίος βρίσκεται σε αδύναμη θέση γιατί πώς μπορεί να περιμένεις καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό και πρέπει να στηρίξουμε τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση στην αγορά εργασίας και πώς θα επηρεαστεί από τους στόχους που βάζουμε για τα επόμενα δέκα χρόνια. Σίγουρα η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας είναι η προτεραιότητά μας. Δεν είναι επίμαχο αυτό το θέμα, εννοείται. Όπως επίσης η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Πρέπει να αξιολογήσουμε λοιπόν την κατάσταση στη σύγχρονη αγορά εργασίας και να δούμε τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν στις χώρες μας. Σίγουρα η κατάσταση είναι διαφορετική στις χώρες που έχουν ε, πολύ εργατικό δυναμικό και διαφορετική στις χώρες εκείνες που υπολείπονται σε εργατικό δυναμικό. Άρα πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση και να βρούμε διαφορετικές λύσεις στην κάθε περίπτωση. Για κάθε εργαζόμενο πάντως είναι πολύ σημαντικό να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τον χρόνο που δουλεύει. Είναι χρήσιμο να υπάρχει λύση εξατομικευμένη. Αυτό όμως που είναι τραγικό είναι ότι παραμένει το πρόβλημα άλυτο και δεν έχουμε καταλήξει σε μια γενική λύση. Πρόεδρος, θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι τους προσκεκλημένους μας. Πρώτον, από ό,τι καταλαβαίνω, εσεί θα προσπαθήσετε να καταλήξετε σε μια συμφωνία μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Θέλω να ρωτήσω την Business Europe, ε, αυτό τι είναι, είναι για να κερδίσετε χρόνο. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι η ιδέα της διαπραγμάτευσης αυτής μεταξύ κοινωνικών εταίρων δεν ήταν και πολύ επίκαιρο, δηλαδή οι πιθανότητες να καταλήξετε σε συμφωνία είναι περίπου μηδαμινές, οπότε γιατί το δεχτήκατε αυτό. Και δεύτερον, μιλήσαμε κάποια στιγμή σε μια προσέγγιση ανατομέα, τομεακή. Δεν είναι πια επίκαιρο αυτό το θέμα και για ποιο λόγο. Γιατί έχετε παρετηθεί από ό,τι δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή από αυτό. Λοιπόν, έχουμε ήδη καθυστερήσει κατά πέντε λεπτά, σίγουρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο και εσείς είσαστε πολύ άριθμοι. Παρ' όλα αυτά θα σας δώσω το λόγο, τι να πω, δυόμιση λεπτά ο καθένας, άντε τρία. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Ανδρέας Πέρσον. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σχολιάσω και εγώ κάπως σύντομα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους τους ευρωβουλευτές για τα σχόλιά τους. Θα επικεντρωθώ σε μερικά ζητήματα. Κυρίως σε αυτά τα οποία χειρίστηκα εγώ. Το θέμα των εφημεριών, για παράδειγμα, που είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τους εργοδότες. Ακόμα και αν υπάρχουν και άλλα θέματα αναφέρθηκε ότι ίσως υπάρχουν δυνατότητες για τελική λύση και είναι ζωτική σημασία για μας να βρεθεί μια τέτοια οριστική λύση. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα που θα μπορούσε εδώ κανείς να θίξει. Για το θέμα της αυτοεξαίρεσης, εμείς στη δικιά μας την απάντηση λέμε ότι, κατά τη γνώμη μας, δεν ε, πρέπει να σταματήσει, αλλά αν το θέμα των εφημεριών λυθεί, κατά τη γνώμη μας, θα μπορούσε να μειωθεί η χρήση του opt-out. Σκόπευα να το πω και πριν στην παρουσίασή μου, αλλά επειδή δεν είχα αρκετό χρόνο το παρέλειψα. Όπως επίσης είπα, στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης είπαμε ότι θέλουμε λύσεις ανατομέα. Και να, και τώρα δηλώνουμε υπέρ του να γίνουν διαπραγματεύσεις ανατομέα. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο να βρούμε μια λύση μεταξύ μας. Θα είναι δύσκολο. Ελπίζουμε όμως να προσπαθήσουμε αν μη τι άλλο και ελπίζω κάποια λύση να βρούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λέει πρόεδρος, ο κύριος Ρίσαρ Ευχαριστώ. Για να απαντήσω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είναι σαφές ότι παρά την οδηγία έχουμε 20 εκατομμύρια στην Ευρώπη που δουλεύουν πάνω από 40 ώρες τη βδομάδα. Αυτό είναι απειλή και στην υγεία και για την ασφάλεια και για την καλή ισορροπία ιδιωτικού χρόνου και εργασίας και για την ισότητα των φύλων. Αν εξακολουθήσουμε να έχουμε, επιτρέπουμε μια τέτοια κουλτούρα, αυτό υπονομεύει ε, οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια για την επίτευξη ισότητας των φύλων και ισορροπία ιδιωτικής ζωής εργασίας. Για το opt-out συμφωνούμε για το ότι ένα βασικό στοιχείο είναι οι εφημερίες που έχει σχέση με την αιτία για το opt-out. Αν και πολλές χώρες έχουν εισάγει το opt-out, δεν ξέρουμε σε τι βαθμό χρησιμοποιείται. Και να δούμε λεπτομέρειες για ορισμένες χώρες χρησιμοποιείται πολύ λίγο. Και στο κέντρο βρίσκονται οι εφημερίες. Είναι ρεαλιστικό λοιπόν να συζητάμε την κατάργηση του opt-out αν βρούμε τις αιτίε του. Και αυτό είναι το βασικό ερώτημα για μας. Πώς μπορεί να έχουμε νομοθεσία για υγεία και ασφάλεια αν αυτό επαφείται σε, στην προσωπική επιλογή. Η κυρία Λίλιαν Βολοσίνσκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τρία σημεία. Το opt-out, το είπα και πριν. Υπάρχει τρόπος να μειωθεί η χρήση του. με την παράταση της περίοδου αναφοράς ως προς τους 12 μήνες, όχι με συλλογικές συμβάσεις, αλλά με εθνική νομοθεσία, Φερρυπίν. Δεύτερο σημείο του κυρίου Σέρκας, σε αιτήσια βάση ο χρόνος εργασίας. Το είχε προβλέψει το Κοινοβούλιο στην πρότασή του και στι προηγούμενε διαπραγματεύσει. Χαιρόμαστε γι' αυτό, για το δηλαδή το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη θέση μα. Το δεύτερο, η νομική βάση και η διάσταση υγεία-ασφάλεια. Ναι, αυτή πρέπει να είναι η νομική βάση της οδηγίας. Και πρώτο ζητούμενο είναι να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια του εργαζόμενου. Αλλά έχουμε να λάβουμε υπόψη και τις εξελίξεις στο χρόνο εργασία, πιο ευέλικτε μορφέ εργασίας, την ανάγκη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Τελευταία του κ. Κρίστενσεν. Ποιοι τομεί χρειάζονται παραπάνω από 48 ώρε τη βδομάδα. Δεν είναι θέμα πάνω από ή λιγότερο από 48 ώρες. Το θέμα είναι πώ θα γίνει ο υπολογισμό, ο μέσος υπολογισμό ή τι περίοδο, γιατί υπάρχουν εχμέ παραγωγής, όπου οι επιχειρήσεις χρειάζονται πάνω από 48 ώρες και άλλες φορές περίοδοι που χρειάζονται λιγότερε ώρες. Γι' αυτό θέλουμε όλε οι επιχειρήσει να έχουν ένα μέσο υπολογισμό 40 ώρων σε μια πιο μακρά περίοδο αναφοράς. η κυρία Ουιρμεκ. Ευχαριστώ. Τομιακές διαπραγματεύσεις, οι δύο τομιακές διαπραγματεύσεις. Για μας το E2C, εμείς θέλουμε διατομιακές διαπραγματεύσεις. Γιατί εδώ συζητάμε θέματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους στην Ένωση. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Κύριε Μάν, με ρωτήσετε για το θέμα των φύλων. Θέλουμε ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τα εργασιακά. Και έχουμε και το άθρο 33 στο χάρτη που είναι νομικά δεσμευτικό. Την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε δεν το είχαμε δεσμευτικό. Αν δούμε τα νούμερα έχουμε παραδείγματα όταν, ας πούμε, σε μια οικογένεια γεννιόνται παιδιά, οι άντρες δουλεύουν περισσότερο και οι γυναίκες δουλεύουν λιγότερο. Είναι αυτό μια προαιρετική αύξηση του χρόνου εργασίας του ανδρός και μείωση του χρόνου εργασίας της γυναικός ή όχι. Για την περίοδο αναφοράς Δεν έχουμε την εικόνα από τους εργοδότες για πού χρειάζεται αυτή η επέκταση. Εμείς θεωρούμε ότι η ευελιξία υπάρχει στην οδηγία. Η δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων υπάρχει. Και ας το χρησιμοποιήσουν οι τομείς που το χρειάζονται. Η κυρία Πρέβικα Σμίθ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους ε, ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Όπως το τόνισαν ήδη κάμπος οι ομιλητές, συμφωνούμε και εμείς ότι η βάση της οδηγίας είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στόχος της οδηγίας αυτός πρέπει να είναι. Ταυτόχρονα Θέλουμε αυτά τα στοιχεία της ευελιξίας που υπάρχουν στην οδηγία να παραμείνουν έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να τα εφαρμόσουν Τέθε ένα ερώτημα ότι γίνεται μια προσπάθεια αναθεώρηση της οδηγίας για την ε, ετήσια αναρωτική άδεια και τις εφημερίες και τι έκανε η Κομισιόν στη διαδικασία αναθεώρησης δεν ήταν μόνο αυτά τα θέματα στο τραπέζι και περιέπλεξαν τη συζήτηση διαβρύνοντας το πεδίο της αναθεώρησης της οδηγίας. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε στα θέματα αυτά. Ο κύριος Θέρκας είπε όπου να φροντίσουμε όχι να δημιουργούμε νέα προβλήματα, αλλά να λύνουμε προβλήματα και συμφωνούμε. Εμείς λέμε, αν γίνει ευρία αναθεώρηση υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε πολλές από τις πολλές καλές ρυθμίσεις που πέτυχαν οι κοινωνικοί εταίροι και οι επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο, σε συγκεκριμένα εθνικά σημεία, οι αυτόνομοι εργαζόμενοι κλπ. Αυτά είναι καλύτερα να ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο. σε συμφωνημένη βάση. Επίσης πρέπει να δημιουργούμε γέφυρες. Προσπαθούμε να βρούμε λύση για επίγοντα προβλήματα. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο, δεν μπορώ να σας δώσω ενδείξεις, κυρία Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή. Γιατί η Business Europe τώρα είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων στην πρώτη φάση στις διαβουλεύσεις δεν κλείσαμε την πόρτα. Τώρα, όπως είπε η συνάδελφος, θεωρούμε ότι το θέμα είναι κυρίως των κοινωνικών εταίρων και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Ιδιαίτερα όσον αφορά την μη πληρωμένη αιτήσια άδεια και της εφημερίας. Πρόεδρος, θα ξαναδώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω στην ερώτηση του κύριου Μαν. Σε τι βαθμό είμαστε σοβαροί για τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Κοιτάστε, υπάρχουν διάφορες αναλλακτικές λύσεις στην ανακοίνωσή μας. Εάν οι περισσότεροι από τους κοινωνικούς εταίρους και από τις δύο πλευρές συμφωνούν με κάποια από τις εναλλακτικέ λύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε αυτή την εναλλακτική λύση θα εγκρίνει στην πρότασή της. Είναι δύσκολο πάντα να βρεθεί κοινός τόπος και από τις δύο πλευρές. Στόχος μας δεν είναι να μοιράσουμε στα δύο τα πράγματα. Θέλουμε να υπάρχει σαφήνεια στις διατάξεις. Πάντως είμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν πολύ διαφορετικές ε, τοποθετήσεις από τις δύο πλευρές. Φυσικά και είμαστε υπέρ της διαβούλευσης και τις λαμβάνουμε υπόψη τα συμπεράσματα δηλαδή από τις διαβουλεύσεις στην έκθεσή μας. Πάντως διευκρινίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει αξιολόγηση. Την μελέτη δημοσίευση, η οποία ανατέθηκε σε έναν εξωτερικό σύμβουλο. Η Επιτροπή στη συνέχεια θα υποβάλει την πρότασή της. Τώρα για τις ε, προσφυγές επί παραβάση. Εφόσον δεν υπάρξει αναθεώρηση της οδηγίας, ε, γι' αυτό ξεκινάει η Επιτροπή προσφυγές επί παραβάση για τις χώρες που παραβιάζουν την οδηγία. Ήδη υπάρχουν ε, για διάφορες ε, χώρες μέλη για όλα τα στάδια. Από αιτιολογημένη γνώμη μέχρι τις προσφυγές επί παραβάση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί για ορισμένες. Και παραμένουν και πολλές άλλες ανοιχτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αλλάξει την νομοθεσία τους οι χώρες μέλη. Και γι' αυτό δεν χρειάστηκε να προχωρήσουμε, γιατί άλλαξε νομοθεσία στο μεταξύ των χωρών μελών, όπως γίνεται και με τις, ε, τα ρεπό. Σε μερικές περιπτώσεις είχαμε 80 ώρες τη βδομάδα. Οι διαδικασίε ξεκίνησαν, τα κράτη-μέλη, όπως σα είπα, πολλέ φορέ άλλαξαν την νομοθεσία του, ακριβώ επειδή ξεκίνησε η διαδικασία προσφυγή επί παραβάση. Είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι σε αυτό το σημείο. Επίσης ο κύριος Χιού ρώτησε κάτι δύσκολο. Η Επιτροπή δεν μπορεί να δοκιμάσει το δικαστήριο. Εμεί αυτό που μπορούμε να πούμε είναι κατά πόσο υπάρχει παράβαση όχι. Και ξεκινάμε μια διαδικασία επί παραβάση. Και αυτό μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε. Το opt-out είναι παραδεκτό το θέμα είναι το opt-out που εφαρμόζουν οι χώρες μέλη είναι έτσι όπως αυτό προβλέπετε ή παραβιάζουν τις ρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ε, πρώτη σας ε, παρουσίαση εδώ. Είπαμε, οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες. Οπότε σας εύχομαι Κοινωνική εταίρη. καλή επιτυχία στις διαπραγματεύσεις που θα έχετε τους επόμενους 9 μήνες και ελπίζω να καταλήξετε σε μια συμφωνία όσο γίνεται καλύτερη. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη, συνεπώς, και ερχόμαστε στην έκθεση του κυρίου Πρίντσια Στερόσα για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και έχουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Περιμένω να ε, φύγουν από την αίθουσα οι προσκεκλημένοι μας. Μιλάμε εδώ πέρα για το μέλλον των ε, υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Ποια θα είναι η εξέλιξη. Και αυτό το κάνουμε στα πλαίσια των συνθήκων όσοι έχουν αυτές. Επικουρικότητα υπάρχει εδώ, άρα έχουν μεγάλη ευθύνη οι χώρες μέλη για να καθορίσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να λάβουμε υπόψη μας ποιες είναι οι ανησυχίες αυτών που προσφέρουν τις γενικές αυτές υπηρεσίες και ποιες είναι οι ανησυχίες του κοινού που υποφελείται από αυτές, που τις χρησιμοποιεί. Γι' αυτό και χρειάζονται διαβουλεύσεις και έκανα διαβουλεύσεις με τους διάφορους εταίρους πριν ετοιμάσω την έκθεσή μου. Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα της αναγνώρισης, του ότι οι κοινωνικές υπηρεσίε γενικού συμφέροντος είναι κοινοφελείς υπηρεσίες βάσει του πώς τις ορίζουν οι χώρες μέλη. Ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που έχει περάσει και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ορίζει μερικές από αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος σαν υπηρεσίες οικονομικού συμφέροντος. Άλλες είναι μη οικονομικού συμφέροντος. Οπότε υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός των μη οικονομικών και των οικονομικών. Δηλαδή μη οικονομικού και οικονομικού συμφέροντος κοινωνικές υπηρεσίες πώς ε, τώρα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Δρούν στα πλαίσια της ε, συνθήκης. Και είναι σίγουρα ένας περίπλοκος τομέας. Αυτό που είναι ξεκάθαρο Είναι ξεκάθαρο ότι δρούν μέσα στα πλαίσια μιας οικονομικής κρίσης και όπως λέω και στην έκθεσή μου, η οικονομική κρίση δημιούργησε πρόβλημα σε αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες συνθήκες. Μετά μάλιστα και από την ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Το άρθρο 14 έχει επεκταθεί και μιλάει για την ευθύνη των χωρών μελών στις 26 τουλάχιστον χώρες. Έχουμε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά. Υπάρχει λοιπόν πολλή κίνηση εδώ, πολλές αλλαγές. Είναι δικιά μας ευθύνη να δράξουμε την ευκαιρία αυτή για να διορθώσουμε ό,τι προβλήματα έχουν προκύψει επί τόπου στην προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος με τέτοιο τρόπο ώστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία να βοηθάει για την καλή διεξαγωγή. Έτσι έχω συντάξει την έκθεσή μου με 37 παραγράφους. Παρόλα αυτά έχω 285 τροπολογίες. Είναι δύσκολο να τη συμπυκνώσω σε μια έκθεση που έχει νόημα. Εξάλλου, το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε εδώ ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που να βάλουμε ό,τι θέλουμε, τα πάντα χωρίς ουσία και χωρίς νόημα. Γι' αυτό και προσπαθούμε μέχρι τον Ιούνιο να ετοιμάσουμε κάτι που να έχει νόημα και όχι που να τα λέει όλα και τίποτα. Πολλές από τις προτάσεις, τις τροπολογίες δηλαδή, ζητούν διαγραφή κάποιων παραγράφων. Όλες οι παράγραφοι στην έκθεσή μου όμως έχουν μπει για κάποιο λόγο, αντικατοπτρίζουν μια πραγματικότητα. Αυτές οι προτάσεις διαγραφής διαγράφουν γεγονότα. Δεν είναι πολιτικές ε, δηλώσεις. Εγώ ευχαρίστω να καθίσω με του συντάκτε των τροπολογιών αυτών και να δω ποια είναι η ανησυχία του και τι θέλουν, γιατί θέλουν να διαγραφούν αυτέ οι παράγραφοι. Να δω μήπω μπορώ να καθισχάσω τι ανησυχίε του με κάποιο τρόπο. Εγώ δεν προσπαθώ να επιβάλλω τη δικιά μου την πολιτική άποψη σε αυτό το τομέα. Λέω ότι χρειάζεται μια οδηγία πλαίσιο, μια ρύθμιση βάσει 48. Δεν προτείνω όμως συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Προσπαθώ να εντοπίσω το πού έχουμε πρόβλημα και πώς μπορούμε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Φροντίζοντας και διασφαλίζοντας την ποιότητα στην προσφορά των υπηρεσιών αυτών. Ποιότητα και για αυτούς που δουλεύουν για τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να πω. Θέλω συνένεση, ευρεία συνένεση για ένα θέμα ουσίας. Το επόμενο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ότι έχω και τροπολογίες για προστίκες. Σήμερα δεν θα μπω στις λεπτομέρειες των 285 τροπολογιών. Ελπίζω να μπορέσω να καθίσω με τους συντάκτες και να λύσουμε διάφορα σημεία. Πάντως υπάρχουν προσθήκες που προτείνονται και που μπορώ να δεχτώ και κάποιες τροπολογίες που θέλουν να αντικαταστήσουν τη δικιά μου διατύπωση σε ορισμένες παραγράφους. Αυτά μπορώ να τα δεχτώ σαν προσθήκες. Δέχομαι ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερη διατύπωση σε μερικές περιπτώσεις, οπότε ευχαρίστω να δεχτώ τέτοιες τροπολογίες. Όμως, χρειάζομαι και επεξηγήσεις για ορισμένες τροπολογίες προτείνεται μια τροπολογία για να αφαιρεθεί η μνήμα που γίνεται στο γεγονός ότι οι κοινέ υπηρεσίες γενικού συμφέροντος αποτελούν προστιθέμενη αξία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με Business Europe το έχει πει αυτό και έχουν πει ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι ζωτική σημασία ώστε να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε γιατί να το βγάλω. Αυτός που το προτείνει αυτό να έρθει και να μου εξηγήσει γιατί, ποια είναι η ανησυχία του ίσως να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία και γι' αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε το σημείο αυτό. Σαν παράδειγμα σας το δίνω αυτό τώρα, δεν θα σας μιλήσω για όλες τις τροπολογίες. Πολλές μπορώ να δεχτώ επί της αρχής επίσης, παρόλο που μπορεί να μην μου αρέσει η διατύπωση. Αλλά και εδώ πάλι αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και να βρούμε ένα συμβαστικό κείμενο. Ένα πάντως από τα θέματα τα οποία με απασχολούν είναι όπως σας είπα πριν οι προτάσεις διαγραφής. Διαγραφή για παράδειγμα για την υψηλού επίπεδου Task Force. Ευχαριστώ την κυρία Μπαστός που προσφέρει και μια εναλλακτική ιδέα για το παρατηρητήριο. Εγώ δεν κολλάω στη γλώσσα, όπως και αν το ονομάσουμε εγώ λέω task force, γιατί θέλω να δείξω ότι είναι κάτι δυναμικό. Αλλά αυτό συζητιέται. Το πραγματικό ζήτημα είναι πώς θα προχωρήσουμε από εδώ που βρισκόμαστε στη συζήτηση αυτού του θέματος στο να πετύχουμε συγκεκριμένη πρόοδο υπέρ των πολιτών μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει Ε, να φροντίσουμε γι' αυτό μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Μα είχαμε εδώ σήμερα το πρωί τον νέο πρόεδρο. Και από ό,τι φαίνεται δεν βοηθάει. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας μας το ξεκαθάρισε σήμερα το πρωί ότι είναι συμβουλευτικό σώμα. Εκπροσωπούνται εκεί οι 27 χώρες μέλη συν η Επιτροπή, χωρίς να είναι όμως πολιτικό σώμα. Οπότε είτε μιλήσουμε για παρατηρητήριο, είτε μιλήσουμε για task force, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σώμα που είναι πολιτικό και ας είναι μικρό, που να μπορεί να πετύχει συνένεση και να πιέσει για αλλαγέ. Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας δεν είναι το κατάλληλο σώμα για αυτή τη δουλειά. Μπορεί να έχει κάποιο ρόλο να παίξει, δεν λέω, γι' αυτό το παρατηρητήριο ή task force όπως και το ονομάσουμε μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο. Αλλά συμβουλευτικά. Είναι διαφορετικό αυτό που ψάχνω εγώ να πετύχω, που θέλω να πετύχω. Αυτά εισαγωγικά για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Μπορώ να προτείνω σε 10 μέρες μια συμβιβαστική πρόταση για να δω αν συμφωνούν οι διάφοροι συντάκτες. Να καθίσω να δω μετά με τους σκιώδεις εισηγητές ποια είναι η απόψή του για το συμβαστικό αυτό κείμενο που θα προτείνω. Έχουμε 4 με πέντε εβδομάδες αν δεν απατώμε πριν επανέλθουμε και ξανασυζητήσουμε. Σε έξι εβδομάδες ψηφίζουμε νομίζω και σε 4 πεντε εβδομάδες θα συζητήσουμε για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ η κυρία Ντελή και η κυρία Μπαστός. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρο, κύριε Σιγητά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά διακυβευόμενα εδώ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και πλήρη επιπτώσεων και είναι ένα συναρπαστικό θέμα γιατί αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε σε ένα χώρο που είναι και τεχνικός αλλά με πολιτικές πτυχές. Είναι ένας πολύπλοκος τομέας στον οποίο πρέπει να, να δράσουμε γιατί οι υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να αντιμετωπιστούμε ένα τέτοιο τρόπο στην Ευρώπη ώστε να οδηγήσει, που να οδηγήσει στην βελτίωσή του. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα κείμενο που να εμφορείται από θελησιοκρατία. Ζητούμε από την, την Κομισιόν να μα προτείνει κάτι περισσότερο, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο επίπεδο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και την κοινωνική πρόοδο. 23 Μαρτίου η Κομισιόν μας έδειξε ότι είχε κατανοήσει αυτό το μήνυμα. Γιατί το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών περνάει κατά ανάγκη από την ε, αρχή κλειδί ότι είναι απαραίτητη η διευκρίνηση και η απλοποίηση των κανόνων, η αναλογικότητα και μια διαφοροποίηση όπως απαιτείται. Ελπίζω λοιπόν κυρία Ισηγητά ότι οι προτάσεις τροπολογίας μου που ο στόχος τους είναι να είναι επικοδομητικές θα ληφθούν υπόψη σας. Ιδίως η τροπολογία μου 119 που προτείνει ένα ταμείο για την κοινωνική καινοτομία και η 169 που έχει να κάνει με τον έλεγχο των υπερβολικών τιμολογίων και επίσης για τον έλεγχο του, μια αντίστοιχη τροπολογία για τον έλεγχο του αριθμού του προσωπικού. Σας ευχαριστώ πολύ η Ριζίνα Μπάστο και μετά η Μαρία Χάρκιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον πρώην CSD Ρώσα, για το έργο που έχει φέρει σε πέρα. Είναι ένα έργο το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αυτό το θέμα δεν είναι ένα θέμα χωρίς ε, ε, πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε, η πολλαπλότητα των τροπολογιών που είχαν παρουσιαστεί στην προηγούμενη έκθεση Φερέιρα που ήταν 285 των αριθμών κατέδειξε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα εξακολουθεί να είναι αντικείμενο έντονων συζητήσεων και φυσικά ένα θέμα το οποίο δεν έχει ε, αποκομίσει μια γενική συνένεση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις ε, αμφισημίες και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι πρέπει να, να παρθούν κάποιες αποφάσεις οι οποίες έχουν ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα. Οι τροπολογίες αυτές οι οποίες έχουν κατατεθεί λοιπόν έχουν ε, σαφώς πολιτικό χαρακτήρα. Η, θέληση του εισηγητή βέβαια δεν είναι να οδηγήσει σε ιδεολογική αντιπαράθεση αυτή την έκθεση και να διχαστεί το Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες είναι τροπολογίες διαγραφής. Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες ζητούν μία αντιμετώπιση η οποία βασίζεται σε προκαταλήψεις. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας. Εγώ κατέθεσα τροπολογίες και άλλοι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καταθέσαμε ορισμένε τροπολογίες διαγραφικού χαρακτήρα. Αυτό δεν είχε σαν στόχο να οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις. Εμείς εμφορούμεθα από ένα πνεύμα συμβιβασμού και θέλουμε να γίνουν οι απαραίτητες διμερείς επαφές για να εξετάσουμε καλύτερα τις τροπολογίες και να θεωρηθούν αυτές οι τροπολογίες ότι είναι θετικές συμβολές για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και σίγουρα σεβόμαστε αυτό το οποίο θέλει ο εισηγητής να μην υπάρξει ένα, ένας εσωτερικός διχασμός του Κοινοβουλίου για ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινωνική συνοχή σε μια οικονομική συνοχή. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν οι τροπολογίες τις οποίες εγώ κατέθεσα εμφορούνται από το πνεύμα της αποσαφήνισης του γεγονότος ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών, ότι η εγκύτητα προς τον πολίτη και τον καταναλωτή έχει τη μεγαλύτερη σημασία και ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινωνικού οικονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους, οι οικομενικές να διέπονται από ένα αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης των πόρων που εξασφαλίζει την ε, ισορροπία, τη συνέχιση αυτής της υπηρεσίας και την προσβασιμότητα σε βασικές υπηρεσίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε τονίσει από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, ότι αυτές οι υπηρεσίες έχουν θεμελιώδη χαρακτήρα. Και επειδή είναι θεμελιώδες, πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία και τη σωστή Να Δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή τώρα να σκεφτούμε να προχωρήσουμε σε περισσότερη ε, ευρωπαϊκή αντιμετώπιση αυτών των υπηρεσιών. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι για μας ακόμα και για την ίδια τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη την κοινωνική πτυχή, είναι απαραίτητο να υπάρχει και μια διευκρίνηση του τι είναι ακριβώς οι υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, είτε είναι οικονομικού είτε μη οικονομικού χαρακτήρα. Έχουμε καταθέσει λοιπόν τροπολογίε προ την κατεύθυνση αυτή. Αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι για μια ακόμα φορά <clears throat> να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι υπηρεσίε θα πρέπει να διευκρινιστεί ο χαρακτήρας τους χωρίς με την επιφύλαξη του να εξασφαλιστεί η σωστή αρμοδιότητα πάνω σε αυτές τις υπηρεσίες που πρέπει να είναι στο εγκύτερο δυνατό επίπεδο για είναι τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές. Έχει προταθεί να υπάρξει ένα παρατηρητήριο το οποίο θα δώσει εναλλακτικέ λύσεις και προτάσεις σε σχέση με την ομάδα υψηλού επίπεδου και αυτή η πρόταση του παρατηρητήριου θα ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο εκκίνησης μετά την ψήφιση αυτής της έκθεσης ως το επόμενο βήμα για την υλοποίηση αυτών των αρχών. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να υπάρξει μια παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος στην Ευρώπη στα κράτη-μέλη που να γίνεται σε επίπεδο περιφερειακών και τοπικών αρχών και επίσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητο να μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία, να έχουμε κατάλογο βελτίστων πρακτικών που μπορούν να είναι συγκρίσιμε, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προ την σωστή κατεύθυνση. Και αυτή <clears throat> η σωστή λοιπόν κατεύθυνση είναι αυτή που μα ενδιαφέρει μέσα από την πρόταση την εναλλακτική τη δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου για τι υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντος. Κλείνω λέγον στον κύριο πρώην σα, στον εισηγητή, ότι είμαι στη διάθεσή του για να συζητήσουμε διμερώς τις προτάσεις αυτές και θα ήθελα να παρακινήσω τον εισηγητή να μην κρατήσει κλειστό πνεύμα σε μια θέση άρνησης προτάσεων διαγραφής ορισμένων παραγραφών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ανοχή σας ό,τι αφορά την υπέρβαση του χρόνου. Α, νομίζω ότι είσαστε στο πνεύμα του εισηγητή. Η κυρία Χαρκίν και μετά η κυρία Λίνκεβιτσιού Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη και ο Στιώδης είναι απόν, θα κάνω τα σχόλια εξ ονόματός του. Καταρχήν ένα γενικό σχόλιο. Οι 250 τόσες τροπολογίες δείχνουν ενδιαφέρον, αλλά δείχνουν και πολιτικές διαφορές. Επειδή ξέρω τον εισηγητή, είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρει να πετύχει συμφωνία. Μερικά σχόλια από το σκιώδη μας. Όλοι συμφωνούμε για την άγνοια να ξεκαθαρίσουν οι κανόνες, αλλά υπάρχουν διαφορές ως προς τις λύσεις. Στόχος είναι να έχουμε την επικουρικότητα με την ευθύνη ότι η Ένωση και οι κυβερνήσεις έχουν σε σχέση με τις αρμοδιότητές τους. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας κατά πόσον ένα νομικό, νομοθετικό πλαίσιο είναι η λύση άλλα σημαντικά θέματα. Στην πρώτη παράγραφο μπορεί να υπάρξει συμβασμός εύκολα σε θέματα ορισμού, ε, ο ενιαίος χαρακτήρας κλπ. Μερικές παράγραφοι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, όπως η 7, η μεγιστοποίηση του κέρδους σε σχέση με την αρχή του SSGI. Στην παράγραφο F είναι δυνατόν να υπάρξει συμβασμό, συγγνώμη 9 και την παράγραφο 10. Η 11 θα είναι μάλλον προβληματική μεταξύ αυτών που θέλει να ενισχυθεί ο προπολογισμό και άλλοι που είναι κατά. Το ίδιο και την παράγραφο 13. Υπάρχει διαφορά. Συμβασμό μπορεί να υπάρξει για την παράγραφο 16, ευρωπαϊκό καθεστώ για τι ε, εταιρείε αμοιβαίου χαρακτήρα. Παράγραφος 17 κρατικές ενισχύσεις, κανόνες προμηθειών, κανόνες Μόντι, Κρόλς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη οι νέες ανακοινώσεις της Κομισιόν. Να αυξηθεί το κατόφλι και οι κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες. Όπως επίσης και ο εξυγχρονισμός των κανόνων. Παράγραφος 18. Υπάρχει δυνατότητα συμβασμού τα κριτήρια στην ταξινόμηση μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών υπηρεσιών δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να βελτιωθούν οι κανόνες, να έχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίε. Και τέλος, μπορούμε να συμφωνήσουμε για την Task Force όσον αφορά την εντολή, του στόχους και τη συμμετοχή. Με δύο λόγια, υπάρχει δυνατότητα βελτιώσεων και πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθούν ορισμένοι συμβασμοί. Βιτσούτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντερόσα. για την πολύ σημαντική δουλειά του. Σας εύχομαι καλή τύχη στους συμβιβασμούς και ελπίζω να εγκριθεί η έκθεση. Οι δικές μου τροπολογίες συμπληρώνουν μερικούς όρους της έκθεσης. Δεν θέλω να περιοριστούμε μόνο στις κοινωνικές υπηρεσίες. Θέλω όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να μπουν μέσα. Έχουμε οικονομικές και μη οικονομικές υπηρεσίες, την εφαρμογή της εσωτερικής μεθόδου στο θετικό δίκαιο της Ένωσης. Ξέρουμε ότι οι αποφάσεις του Ευρωδικαστηρίου δεν αρκούν για να έχουμε νομική βεβαιότητα και για την παροχή των υπηρεσιών αυτών από, τα, από φορείς. Έχω και μια τροπολογία για τη φύση των υπηρεσιών αυτών. Καταρχήν λέμε ότι είναι πολύ ειδικού χαρακτήρα αυτές οι υπηρεσίες είτε αναφέρονται σε άτομα με ειδικέ ανάγκες. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι αυτοί που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες είναι και αυτοί ειδική μορφής. Πολύ συχνά είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, ε, οργανώσει που δουλεύουν σε εθελοντική βάση, άτομα, επιμέρους. Ο ειδικό χαρακτήρας λοιπόν αυτών που παρέχουν αυτέ τις υπηρεσίε έχει σχέση με το ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τη λογική της αγοράς. Δεν δουλεύουν για κέρδος. Και ό,τι ώρες και να ορίσουμε για τη δραστηριότητά τους, οι υπηρεσίες αυτές εξαρτώνται από τη δουλειά των ανθρώπων και όχι από τους όρους. Αυτοί που δουλεύουν στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών θα πρέπει να υποστηριχθούν διότι η φήμη και οι συνθήκες εργασίας πρέπει να βελτιωθούν. Είναι μόνος τρόπος για να τραβήξει κανεί άτομα να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Η ανάγκη για τις κοινωνικές υπηρεσίες στο μέλλον θα αυξηθούν και λόγω δημογραφικών αλλαγών και λόγω εξελίξεων στην κοινωνία. Και εύχομαι κάθε τύχη στον εισηγητή, γιατί πρόκειται για μια τεράστια δουλειά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ο εισηγητής και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στη συζήτηση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω επίσης όλους ότι είμαι απόλυτα έτοιμος να προχωρήσω σε συμφωνία και να συζητήσω μαζί σας. Θέλω να έχω μια ευρεία συνένεση. Αλλά σίγουρα υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να πετύχει κανείς μια ευρεία συνένεση. Μπορεί να καταλήξει κανείς με μια συνένεση καινή περιεχομένου. Επειδή βάση αυτό που άκουσα σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να καταλήξει αυτή η Επιτροπή σε μια έκθεση η οποία περιέχει προστιθέμενη αξία για αυτούς οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος στα κράτη-μέλη και που οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν τη συζήτηση και να προβάλλουν αλλαγές που μπορούν να λάβουν χώρα. Είναι έκθεση πρωτοβουλία, όχι νομοθετικού χαρακτήρα. Ελπίζουμε ότι θα έχει κάποια επιρροή στον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν αυτέ οι υπηρεσίε. Και εγώ δεν θέλω να αποκλείσω τη συζήτηση. Χαίρομαι τη συζήτηση. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε κάποια συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων σε αυτή τη συζήτηση και στο Κοινοβούλιο γενικά είναι περισσότερη συζήτηση και γι' αυτό θέλω από ένα πρώιμο στάδιο να παρουσιάσω ένα σχέδιο συμβιβαστικών τροπολογιών που μπορούν στη συνέχεια και οι να επεξεργαστούν και να επανέλθουν σε μένα και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι. Δεν ξέρω αν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στο στάδιο αυτό εκτός από το να πω ότι χαίρομαι με την απάντηση που δόθηκε για τα θέματα αυτά, για την απόκριση των συναδέλφων. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι αυτή η έκθεση δεν μπορεί να εγκριθεί. Φυσικά θα μπορέσει να εγκριθεί ως συνολικό έργο των μελών αυτής της Επιτροπής. Μπορούμε με την συνεργασία μας να επιτύχουμε μια καλύτερη έκθεση και εγώ ως, αν θέλετε, διαμεσολαβητής μεταξύ των διαφόρων απόψεων. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω να επιτύχουμε κάτι τέτοιο μέχρι τη στιγμή που θα έρθουμε πίσω το Μάιο να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιγητά, λέει η Πρόεδρος. Έχετε ένα μήνα πάνω από ένα μήνα μπροστά σα για να μπορέσετε να διαπραγματευτείτε αυτή την τόσο ωραία συμβιβαστική λύση που στις 24 Μαου θα συζητήσουμε ασμένω για να την ψηφίσουμε στι 25 την επαύριον αυτή τη ημέρα. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση του κυρίου Κώσσα για την κινητικότητα και τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες και τη στρατηγική, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2010-2010 πρόκειται για την εξέταση του σχεδίου ε, έκθεσή σας και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή γιατί και εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο ζει με αναπηρίες όπως βλέπετε και γιατί η έκθεση η οποία μας απασχολεί έχει σαν στόχο να καλύψει τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι με υποστήριξαν σε αυτή την, ε, την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω τη βοήθεια που πήρα για να έχω μια καλή εικόνα των θέσεών σας για αυτή την έκθεση που θέλω να σας παρουσιάσω εν συντομία στις κύριες ε, γραμμές της. Μια θεμελιώδης έννοια στην έκθεση αυτή είναι ότι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό που προσπαθεί να επιτύχει η έκθεση, θα πρέπει να υπάρξει βιωσιμότητα στα μέτρα, θα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικότητα σε όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε μία εφαρμογή της σύμβασης και του πρωτοκόλου που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τα άτομα με αναπηρίες που δεν επαρκούν όμως αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να υπάρξει και μια στρατηγική για το 2020 και η στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία να επιτρέψουν να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή σε ίση συνθήκη με αναπηρία. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό σε νομοθετικό επίπεδο και έχουμε μια σειρά από δομικά θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει μια Ευρώπη χωρίς καθόλου φράγμους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης ότι τα άτομα με αναπηρίες ως κοινωνική ομάδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μέσα στο γενικό κατάλογο των ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες και να εφαρμόζεται να εφαρμόζεται πλήρως η νομοθεσία στα θέματα αυτά. Αυτά είναι τα σημεία ε, εκκίνησης της έκθεσης αυτής. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και συνεκτικότητα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές στρατηγικές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μία σειρά από μέρημνες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Καταρχήν η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων με αναπηρίες. Υπάρχουν πάνω από 80 εκατομμύρια αναπήρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασής τους στην εργασία. Θα πρέπει να καταργηθούν οι διακρίσεις που ισχύουν έναντι των ατόμων αυτών θα πρέπει να γίνει δυνατό <clears throat> τα άτομα αυτά να έχουν καλύτερη ε, πρόσβαση στις επικοινωνίες και τις μεταφορές. Χρειαζόμαστε και καλύτερη συλλογή στοιχείων σε σχέση με τα άτομα αυτά και πρέπει να εξασφαλίσουμε περαιτέρω την ισότητα ευκαιριών για τα άτομα αυτά και να λάβουμε υπόψη μας και τις δημογραφικές ε, εξελίξεις και να εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα των ατόμων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χώροι θα πρέπει να είναι ε, προσβάσιμοι και σε άτομα ηλικιωμένα. Θα πρέπει γενικά λοιπόν να επενδύσουμε περισσότερο για τα άτομα με αναπηρία στο μέλλον και κάτι ακόμα που είναι απαραίτητο είναι να αντιμετωπίσουμε την ένδια που πλήττει πολλά από αυτά τα άτομα και επομένως να βοηθήσουμε τους αναπήρους γιατί μεταξύ των αναπήρων είναι πιο μεγάλο το ποσοστό των ενδεών. Θέλω να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παρέμβει πολλές φορές υπέρ των ατόμων με αναπηρίες. Υπάρχουν πολλά ψηφίσματα τα οποία έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ψηφίσματα αυτά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι απετελέσαν τη βάση για την εκθεσή μου και μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά μέσα σε αυτές τις εκθέσεις Θέλω να είμαι, σε αυτήν την έκθεση θέλω να είμαι πιο αποφασιστικός, διεκδικώντας πιο έντονες παρεμβάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι ε, υπεύθυνο και για μια μη κυβερνητική οργάνωση και δίδω μεγάλη σημασία στη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα αυτό και στις 30 Μαρτίου θα προχωρήσω σε έντονες διαβουλεύσεις με μια σειρά από μη κυβερνητικές προχώρησα συγγνώμη, σε μια έντονη διαβούλευση με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις και είχα πολλές θετικές πληροφορίες που πήρα αυτές και χαίρομαι και για την, ε, τις καλές επαφές που είχα με τους χειώδες εισηγητές οι οποίοι έδειξαν την ε, συνένεσή, της, τους για να ενσωματώσουμε και τις γνώμες, τι γνωμοδοτήσει των μη κυβερνητικών οργανώσεων μέσα στην έκθεση αυτή, εμπλουτίζοντας έτσι την έκθεση. Πιστεύω λοιπόν ότι με όλα αυτά τα στοιχεία προ το τέλο Ιουνίου η έκθεση αυτή θα έχει, μετα... θα έχει βελτιωθεί, θα έχει ε, βελτιστοποιηθεί και θα μπορούμε να έχουμε την υποστήριξη από όλε τι πολιτικέ ομάδε για τα άτομα με αναπηρία και βασίζομαι σε εσά, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Λίνκεβιτσιούτε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια στην ομάδα των σοσιαλιστών. Καταρχήν ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, καλό προετοιμασμένο κείμενο και για την θετική συνεργασία που είχαμε. Συναντηθήκαμε κάποιες φορές, συζητήσαμε το σχέδιο έκθεσης. Ο εισηγητής τόνισε τη σημασία της αύξησης της κινητικότητας άτομα με αναπηρίες, την ανάγκη να έρθουν όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες και θα πρέπει να εφαρμόσουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία και σε εθνικό επίπεδο. Τώρα μερικά σχόλια. Τα κύρια εμπόδια στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία είναι η υψηλή ανεργία. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν είναι καλά προετοιμασμένοι για να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Έπειτα όταν τα άτομα και παιδιά με αναπηρίες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία γιατί η διδακτέα ύλη δεν είναι προσαρμοσμένη ειδικά για τα άτομα αυτά και τα σχολεία τα ίδια δεν είναι προσαρμοσμένα. Αυτό είναι μια, ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους τα άτομα με αναπηρίες υποφέρουν από αποκλεισμό. Κάθε χώρα θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση ε, όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας και θα πρέπει να εφαρμοστούν ενεργές πολιτικές συστήματα που θα ενθαρρύνουν τα άτομα με αναπηρίες να εργάζονται και οι εργοδότες να έχουν κίνητρα να δημιουργούν απασχόληση για άτομα με αναπηρίες. Πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθετική βάση. Επίσης, έχουμε το ότι ακόμα δεν έχουμε ε, έναν θεσμό κάποιο ο οποίος θα βοηθάει τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Ένα τέτοιο θεσμό θα βοηθούσε τους ε, τυφλούς, τους κοφούς να βρούνε τη θέση τους στο χώρο εργασίας. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τις κυβερνήσεις τις αναπηρίες να μην τι αντιμετωπίζουν σαν ένα σωματικό πρόβλημα, περισσότερο να βλέπουν την κοινωνική πτυχή των αναπηριών. Άτομα δύο άτομα που έχουν την ίδια αναπηρία μπορεί να έχουν διαφορετικό καθεστώς, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές δυνατότητες. Ο ένας μπορεί να δουλεύει στην Ήπεθρο και να μην μπορεί να έχει κοινωνικές υπηρεσίες, άρα κοινωνικά είναι αποκλεισμένο. Χάνει δικαιώματα. Πληροφορίες και βοήθεια πρέπει να δίδεται σε οικογένειες που έχουν παιδιά με αναπηρίες και θα πρέπει να περάσουμε από την φροντίδα που παρέχεται από εξειδικευμένα ιδρύματα σε περίθαλψη και φροντίδα που να παρέχεται από την κοινότητα. Χρειάζονται διαρθρωτικά κονδύλια και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν νέα υποδομή να προσαρμοστεί ε, για αυτούς που εκπαιδεύουν, για αυτούς που εφαρμόζουν τα μέτρα κοινωνικής περίθαλψης, σωστούς κανόνες εργασίας, υποστήριξη των οικογενειών και των συγγενών. Σωστή, ε, σωστή περίθαλψη υγείας για άτομα που ζουν και που εργάζονται μέσα σε ειδικά ιδρύματα, σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων με αναπηρίες και ένα πιο συγκεκριμένο πρόβλημα τώρα, η πολιτική ενσωμάτωση που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη διαφέρει από χώρα σε χώρα. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αλλά η διαδικασία ενοποίησης δεν προχωράει πολύ. Συχνά ασχολούμαστε με τις συνέπειες του αποκλεισμού και όχι τις αιτίε. Καταρχήν πρέπει να αρθούν τα εμπόδια. Να δούμε τι οδηγεί σε προβλήματα αποκλεισμού, ανεργίας κλπ. Και τελειώνουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. από τους τυφλούς, από την Ένωση Τυφλών. Υπάρχει ένα, ένα όργανο, Mean Europe λέγεται, στις Βρυξέλλες για τους τυφλούς. Για αυτούς τα μέτρα με την αφή είναι από τα πιο σημαντικά. Πέρυσι οι τυφλοί μπορούσαν να αγγίζουν τα αντικείμενα σε εκθέματα σε αυτό το συγκεκριμένο πάρκο στις Βρυξέλλες. Φέτος ανακοινώθηκε ότι οι τυφλοί δεν μπορούν να αγγίζουν τα αντικείμενα. Μιλάμε και λέμε για πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Στις Βρυξέλλες μάλιστα, πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, Εγώ ασχολήθηκα πολύ με τα άτομα με αναπηρίες. Ενθάρρυνε την έκθεση αυτή. Φυσικά πρέπει να αποφύγουμε τις παγίδες, να ζητάμε πολλά πράγματα που δεν είναι ρεαλιστικά. Η έκθεση Ανταμκούσα αποφεύγει αυτές τις παγίδες, αποφεύγει τις κοινοτοπίες. αποφεύγει τα συμβατικά και επικεντρώνεται στα κρίσιμα θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, κατάργηση της άγγισης μεταχείρισης, και σημαντικά σημεία όπως η ερμηνεία των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία μια ευκαιρία επένδυσης στο μέλλον. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική υπέρ των ατόμων με αναπηρία και προτείνει χρήσιμα μέτρα. Είναι μια χρήσιμη έκθεση, ρεαλιστική, χωρίς κοινοτοπίες. Σας καλώ να την υποστηρίξουμε. και χαίρομαι γιατί ότι ο συντονισμός με τις άλλες ομάδες είναι πάρα πολύ καλός. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι για την έκθεση αυτή. Τελευταία η κυρία Αρκίν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για την έκθεση αυτή, όπως είπε και ο κύριος Όρη, και έχουν καλυφθεί αυτά τα θέματα. Ήδη η κυρία Λίν που είναι η τη εισηγήτρια ζήτησε να πω ορισμένα λόγια εξ ονόματός της, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα. Χωριστά όμως από αυτά τα θέματα θα ήθελα να κάνω ένα παραπάνω σχόλιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο εισηγητής έχει θέσει το θέμα αυτό στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρώπης του 2020 και εμπλέκεται και στην διαδικασία για ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης για όλους. Και στην παράγραφο 9 κοιτάζει πολύ περισσότερα θέματα που έχουν να κάνουν με την αναπηρία από απλώς την παροχή υπηρεσιών. Νομίζω ότι ένας από τους στόχους μας είναι να μειώσουμε και τον αριθμό των ατόμων σε ένδια, δεδομένου το ότι τα άτομα με αναπηρία είναι πολύ πιο πιθανό να βρίσκονται σε κατάσταση ένδυας από ότι ο γενικός πληθυσμό ίσως θα μπορούσε να υπάρξει δυνατότητα να πάρουμε τα στοιχεία τα οποία να είναι ε, εξειδικευμένα ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες ατόμων, ώστε να ξέρουμε πόσα άτομα τα οποία είναι ανάπηρα είναι και σε ένδια. Επίσης, από την πλευρά της κυρίας Λίν, τα σχόλια της είναι εξής. Είπε ότι η στρατηγική αυτή είναι μια σημαντική πτυχή της ε, προσήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες και να τους δώσει απαραίτητες υπηρεσίες. Ο πληθυσμός σας επίσης γυράσκει και μη διδασκόμενο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτε μα ζουν πολύ περισσότερο και επομένω έχουν και περισσότερα προβλήματα με αναπηρίε. Επομένω, είναι απαραίτητε οι καλύτερε πρακτικέ και η μεταλαμβάνευσή του για να αντιμετωπίσουμε το γεγονό ότι θα έχουμε πιο πολλά άτομα με αναπηρίε στο μέλλον και είναι απαραίτητο αυτή η στρατηγική να γίνει σωστή ώστε να ενισχύσουμε την δέσμευσή μα για ίση μεταχείριση των πολιτών με αναπηρία. Είναι απαραίτητο επίση το γεγονό ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε την πρόοδο που επετέφθη με την προσπογραφή της, συμφωνή, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. 11 κράτη-μέλη δυστυχώς δεν έχουν υπογράψει ακόμα αυτή τη σύμβαση. Χρειάζεται πολιτική θέληση στο Συμβούλιο για να ξεπλοκαριστεί το θέμα της ίσης μεταχείρισης ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίσα δικαιώματα και ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες. Με όλε αυτέ λοιπόν τι παρατηρήσει, εγώ χαιρετίζω την πρόταση τη Κομισιόν, ιδίω με την μνήα τη σύμβαση του ΟΗΕ και τις οδηγίες του 2000 για την ισότητα. Ξέρω ότι υπάρχει η πρόταση από την Κομισιόν μιας ενδεχόμενης πράξης για την προσβασιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά προς το παρόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις προτάσεις οι οποίες ήδη είναι εν εξελίξη, προτού περιμένουμε την υποβολή νέων νομοθετικών μέτρων. Θέλω, θε, τέλος κύριε θέλω να ευχαριστήσει τον κύριο ε, Κόζα και τους συναδέλφους του ομάδα, στη διαπαραταξιακή ομάδα για τα άτομα με αναπηρία. Έχουν παρουσιαστεί ήδη προτάσεις από αυτήν την πλατφόρμα για την πρόταση αυτή και ζητά από τον συγητή να εξετάσει αυτή την ε, τροπολογία και φυσικά και του κοιόδε συγητέ να είναι προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα προτού θέσουν τι δικέ του τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κώστα και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους για τις παρατηρήσεις τους μου επιβεβαιώσατε ότι είμαι στο σωστό δρόμο. Ομολογώ απόλυτα ειλικρινά ότι όταν ξεκίνησα να δουλεύω πάνω στην έκθεση αυτή, είχαμε ε. πάρα πολλές ιδέες, ένα τεράστιο κατάλογο με ιδέες. Και βλέπαμε ήδη από την αρχή ότι έπρεπε να ζητήσουμε και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να συμμετάσχουν. Καταλαβαίναμε από την αρχή ότι δεν ήταν δυνατό να κρατήσουμε ένα τέτοιο μεγάλο κατάλογο με ιδέες. Έπρεπε να προσδιορίσουμε τους στόχους μας και να είμαστε ρεαλιστικοί. Μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή στρατηγική με χρήσιμο τρόπο. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω κάποια παραδείγματα. Όσοι πήραν το λόγο ήδη αναφέρθηκαν στο τι είναι το ουσιαστικό και το τι όχι. Το ουσιαστικό είπαν είναι να γίνονται σεβαστά και να τηρούνται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Γιατί τα άτομα με αναπηρίες έχουν ανάγκη από τον σεβασμό αυτό της κοινωνίας. Μια άλλη ιδέα είναι η συλλογή δεδομένων. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρέμβει όσο δεν διαθέτει αξιόπιστα δεδομένα για τα άτομα με αναπηρίες. Πόσα είναι αυτά σε κάθε χώρα μέλος, για παράδειγμα. Όσο δεν γνωρίζουμε λοιπόν για πόσα άτομα μιλάμε, πόσα άτομα με αναπηρίες ζουν σε κάθε χώρα μέλος, δεν μπορούμε και να τα βοηθήσουμε με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Πιστεύω επίσης ότι οι δημογραφικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρο είναι πολύ σημαντικές. Με την έκθεσή μου επιθυμώ να δείξω ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα είναι πολύ φορτωμένα επειδή τα άτομα με αναπηρίες χρειάζονται πολλών ειδών υπηρεσίες προς όφελός τους. Για μένα έχει μεγάλη σημασία τα διάφορα προϊόντα να είναι στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Οι δημόσιες αγορές έπειτα. Και εδώ δίνω μεγάλη σημασία. Σίγουρα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί επί μακρό. Και κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου προς το παρόν. Πρέπει να επικεντρωθούμε και στον τομέα της απασχόλησης. Η απασχόληση πρέπει να είναι ανοιχτή Συγχρόνω όμως πρέπει να υπάρχει προστασία για τα άτομα με αναπηρίες. Πολλά τέτοια άτομα δεν θα μπορέσουν ποτέ να συμμετάσχουν στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να εξασφαλίσουμε και για αυτά τα άτομα κάποιες θέσεις απασχόλησης. Επίσης πρέπει να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι συνάδελφοι είπαν ότι είναι σημαντικό οι φοιτητέ με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες σε όλες τις χώρες μέλη. Να μην γίνονται διακρίσεις. Αυτό όμως είναι αρμοδιότητα του κάθε πανεπιστημίου. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Επενδύοντας στα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα αυτά θα γίνουν ανταγωνιστικά και θα μπορέσουν έτσι να δουλέψουν, θα πληρώνουν φόρους και οι φόροι αυτοί θα αποτελούν την επιστροφή, δηλαδή την αποζημίωση κατά κάποιο τρόπο που θα προσφέρουν τα άτομα αυτά στο κράτος για αυτά που έχει επενδύσει αυτό για εκείνους. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας, για τις παρεμβάσεις σας και περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τροπολογίες σας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να καταλήξουμε σε μια ευφυή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. κύριε Κάζα, για το σχέδιο έκθεσή σας, το οποίο θα είναι αντικείμενο τροπολογιών μέχρι, μέχρι τις 27 Απριλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, το μεσημέρι. και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό στις 24 Μαΐου για να υπάρξει η έγκρισή τους <clears throat> αφού πάρουμε και τις ε, γνωμοδοτήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος, ε, Αναφορών και άλλων. Θα ήθελα τώρα μετά από αυτό το σημείο, πριν φτάσουμε στο σημείο 20, να σας πω για τον τριγωνικό διάλογο, ο οποίος έλαβε χώρα χθες σε σχέση με την έκθεση Κάστλα που αφορά το ευρωπαϊκό έτος της ενεργούς γύρενσης. Ο πρώτος ψυχολογικός διάλογος δεν οδήγησε σε καρπούς και στο πέρας των διαπραγματεύσεων μας επέτρεψε όμως να προχωρήσουμε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό κέριων σημείων και ακολουθούσε τις επιθυμίες της Επιτροπής μας στη ψηφοφορία, παραδείγματος χάρη την έννοια της εισαγωγής μιας κουλτούρας ενεργούς γύρανσης. Το δέχτηκε το Συμβούλιο. Και επίσης εισήχθη η έννοια της πολυμορφίας και της μη διάκρισης κατά τη διάρκεια της ενεργούς γύρανσης. Επίσης επιτύχαμε μια συμφωνία σε σχέση με τον ορισμό αυτών που θα πρέπει να παρέμβουν ε, στο έτος αυτό ε, ενεργούς γύρανσης που να περιλαμβάνει εταίρους από τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μας παραμένει μονάχα τώρα στα πλαίσια του επομένου τριγωνικού διαλόγου του, της 3ης Μαΐου να αντιμετωπίσουμε δύο θέματα τα οποία είναι ακαθόδη, αλλά ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Πριν από το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας, για να περατωθεί η πρώτη ανάγνωση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα του τίτλου της έκθεσης και της γραμμής του προϋπολογισμού που είναι ο διάβολος υποκρύπτων εαυτών εν, τις λεπτο, λεπτομερίες. Μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στο σημείο 20 που θα με κάνει εμένα την ίδια να παρουσιάσω το ειδικό μου ίδιο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 και αυτά τα οποία θα πρέπει να είναι ο καθορισμός της εντολής της Επιτροπής Προϋπολογισμών για τον τριγωνικό διάλογο για τις αρμοδιότητες δικής μας Επιτροπής. Σας υπενθυμίζω ότι η συγγήτριά μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών αυτή τη χρονιά η κυρία Φραντσέσκα Μπαλτσάνη και η γνωμοδότηση την οποία προτείνω εδώ περιλαμβάνει τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας για τη διαδικασία προπολογισμού του 2012, όπως έχουν εγκριθεί από τους συντονιστές κατά την διάρκεια μίας συνάντησης της 10ης Μαρτίου του ενεστώτος έτους. Το ίδιο αυτό περιεχόμενο της γνωμοδότησης συμπεριλαμβάνει και το γενικό πλαίσιο ως οικός μέσα στο οποίο πρέπει να εγγράφει το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την στρατηγική 20 αλλά και 20 η οποία εμπλέκει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας από δύο πτυχές, δηλαδή σε σχέση με δύο στόχους, από τη μία πλευρά αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και δεύτερον αγώνας κατά της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού και επίσης και από τις τρεις πρωτοβουλίες φάρους, νέες, πρωτο, νέες προικανότητες για νέες απασχολη, απασχολήσεις και αγώνα κατά της ένδυας. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι ο προϋπολογισμός των κρατών μελών να είναι αναγνώσιμος εν συμπληρωματικότητα με τον υπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την πλήρη υλοποίηση αυτής της στρατηγικής 2020, προτείνουμε επιπλέον να υπογραμμίσουμε την σημασία που επέχει η ύπαρξη καινοτόμων πόρων και αποτελεσματικών πόρων που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση των κονδυλίων του κοινωνικού τομέα θέλουμε να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε όπως κάναμε και χθες το θέμα της αναδιάθρωσης των επιχειρήσεων και της πρωτοβουλία η οποία θα πρέπει να αναλυθεί προς την κατεύθυνση αυτή εν τέλει στους τομείς που υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές του προπολογισμού, Ταμείο Προσαρμογής στην ε, παγκοσμιοποίηση, το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κτλ. Ζητούμε από τις αρχές, από τους σταγούς του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξασφαλίσουν ότι αυτές οι γραμμές του προϋπολογισμού θα τύχουν πλήρης χρηματοδότηση και θα χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες ευμενής ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Τελευταίο σημείο το οποίο αποτελεί μια προσθήκη και μας φάνηκε απαραίτητο λόγο του νέου πολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο εγγράφεται ο προϋπολογισμός του 2012 είναι η λήψη υπόψη της εταιρικότητος με την νότια όχθη της Μεσογείου που είναι στα σπάργανα αυτής. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή σε αυτή την εταιρική σχέση για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του κοινωνικού διαλόγου και την έγκα δίδρυση και περαιτέρω ανάπτυξη μιας εταιρική σχέσης σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει ένα κλίμα έφορο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και εδώ θα πρέπει να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτέ είναι οι γενικέ κατευθύνσει που θα σα δώσω στα πλαίσια αυτή τη γνωμοδότηση. Αλλά βλέπω ότι η κυρία Τουρούνεν όπω και η κυρία Αρκίν θέλουν να παρέμβουν. Ο πρώτη κυρία Τουρούνεν έχει τον λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ δύσκολο να μη συμφωνήσει κανείς με αυτήν την πρόταση. Είναι μια πολύ καλή πρόταση. Το πρώτο σημείο υπογραμμίζει ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τη στρατηγική για το 2020. Η στρατηγική αυτή δεν έχει χρηματοδότηση ακόμα, άρα πρέπει να έχει αν θέλουμε να πετύχει τους στόχους της. Δεύτερον, το σημείο 10 για την Βόρεια Αφρική είναι επίσης πολύ σημαντικό και είναι πολύ ενδιαφέρον που το φέρνετε εδώ στην Επιτροπή μας. θα υποβάλουμε μια τροπολογία για να επεκταθεί περισσότερο το σημείο 8 που αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε πλήρως δηλαδή το ταμείο αυτό για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης όσον αφορά την νεότητα και την εκπαίδευση. Χωρίς να αλλάξουμε το περιεχόμενο, να επεκταθεί περισσότερο. Έπειτα, σκέφτομαι μήπως μπορούμε να προσθέσουμε ένα σημείο, δεν ξέρω βέβαια αν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, αλλά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι όταν υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε και το θέμα των νέων πόρων, νέων πηγών προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η επαγγελματική κατάρτιση κλπ. Δεν ξέρω αν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, μπορούμε να το συζητήσουμε πάντως για να δούμε. Η προθεσμία είναι το Μάιο, αν δεν απατώμε. Οπότε έχουμε, νομίζω, χρόνο. Πάντως συμφωνούμε απόλυτα με αυτή την καλή γνωμοδότηση. Πρόεδρος. Η κυρία Χάρκιν και μετά ο κύριος Θερκάς. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την προλαλή σας. Κύριε Συγκήτρια, πράγματι, καλύψατε τα κύρια σημεία που θέλει η Επιτροπή μας να συμπεριληφθούν. Έχω όμως κάνα δύο σχόλια. Στην παράγραφο 4 λέτε ότι αν οι πόροι που διατίθεται δεν χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο περισσότερο καινοτόμο και αποτελεσματικό, τότε η δημοσιονομική εξυγένση των κρατών μελών δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Ναι, αλλά πώς, χρειάζεται κάποια καινοτομία εδώ. όταν λέτε ότι δεν υπάρχει συμβατότητα ή συμπληρωματικότητα, είναι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα κράτη-μέλη που δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλλά βέβαια καταλαβαίνω την πρόθεσή σας και συμφωνώ με αυτή. Έπειτα για τις μακροοικονομικές ε, διευκολύνσεις στο σημείο 7. Το στηρίζω. Θα τόνιζα περισσότερο το ότι μπορεί να βοηθήσει αυτό στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει κλπ. Υπάρχει δηλαδή κάποιο δυναμικό εδώ που πρέπει να φανεί. Επίση, μιλάτε και για το Ταμείο για τι επιπτώσει από την παγκοσμιοποίηση. Και μιλάτε για αναδιαρθρώσει επιχειρήσει, βέλτιστε πρακτικέ κλπ μπορεί και αυτό να επεκταθεί περισσότερο. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά ίσως θα πρέπει να το επεκτείνουμε περισσότερο. Και επειδή είχαμε τη συζήτηση που μόλις είχαμε για την προηγούμενη έκθεση για τα άτομα με αναπηρίες, άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια, συμφωνώ με αυτά που προτείνεται, ότι δηλαδή τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απευθύνονται στους μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι η Ρώμα. Αυτό πρέπει σίγουρα να τονιστεί όλος ιδιαίτερος. Κύριο Θέρκαφ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με κάθε συντομία νομίζω ότι εδώ δεν πρόκειται για να δημιουργήσουμε τις ε, ανάδελτους που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για τις ουσιαστικές, για τις πρωτοβουλίες φάρους, χρειάζεται να υπάρχει μια χρηματοδότηση η οποία να είναι επαρκής. Μια ικανή λοιπόν χρηματοδότηση η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τους απαραίτητους πόρους. ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους στόχους της Ευρώπης 2020. Το επομένω είναι καλύτερο αντί να πούμε επαρκή να πούμε μια ουσιαστική χρηματοδότηση. Λοιπόν, σας προσκαλώ να καταθέσετε τροπολογίες εφόσον το επιθυμείτε. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Θα υλοποιηθούν και θα πάρουν σάρκα και μελάνι σε τροπολογίες από τη δική σας πλευρά. Εγώ από τη δική μου πλευρά Υπήρξε ένα σημείο το οποίο δεν μπόρεσα να το παρουσιάσω λόγω των περιορισμών που έχουμε όλοι μέχρι στιγμής, αλλά θα ήθελα να προκαταλάβω λοιπόν τη συζήτηση σε σχέση με τις διαμεσολαβήσεις που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τη δημιουργία ενδιαμέσων κατηγοριών σε σχέση με το Ταμείο Συνοχής και την ανάγκη Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Εμεί δεν θέλουμε να υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία τα οποία θα αποβούν σε βάρος της χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό μέσα από τροπολογία Σα Ευχαριστώ λοιπόν για τι συνεισφορέ τη συζητησή σα, Προτείνω μια προθεσμία κατάθεση τροπολογιών μέχρι τι 5 Μαΐου, 24 Μαΐου θα συζητήσουμε και στι 25 θα ψηφίσουμε, έχουμε, θα επανέλθουμε 25. Τελευταίο σημείο και ίστατο στη μέση διάταξή μα. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Έντιθ Μπάουερ η οποία ανέμεινε τόσο πολύ χρόνο αλλά οι εργασίες μας ούτως είχαν οργανωθεί. κυρία Μπάουερ, σας δίνω το λόγο για την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησή σας για την απορρόφηση των διαφορετικών πόρων και του Ταμείου Συνοχής και το μέλλον αυτών των πόρων, τα διδάγματα τα οποία πρέπει να αντιλήσουμε. Είναι μια προς την Περιφερειακή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι ε, σύντομη. Και ευχαριστώ τους συναδέρφους που εξακολουθούν και βρίσκονται εδώ. Δέχομαι οποιαδήποτε κριτική έχετε να κάνετε, γιατί πράγματι λείπουν ακόμα αρκετά πράγματα σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ε, ουσιαστικά είναι το ένα τέταρτο το κείμενο που έχετε μπροστά σα από το κείμενο που αρχικά είχα ετοιμάσει, επειδή πρέπει να περιορίζουμε το μέγεθος των γνωμοδοτήσεών μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λοιπόν, θα είναι ένα από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την υλοποίηση της στρατηγικής 2020. Δεν είναι σύμπτωση που δίνουμε τόση σημασία στο ταμείο αυτό, λοιπόν, η έκθεση και η γνωμοδότησή μου επικεντρώνεται στα προβλήματα τα οποία περιορίζουν την ε, χρήση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εξυπηρετεί πολλούς ανθρώπους. Θα μπορούσε όμως να είναι ακόμα πιο χρήσιμο. Ένα από τα προβλήματα που εντοπίσαμε στις αναλύσεις που κάναμε είναι ότι υπάρχουν καταστάσεις κατά τις οποίες αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη τα χρήματα αυτά δεν καταφέρουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Στην έκθεση της κυρίας Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ διαβάζουμε ότι το ταμείο αυτό δεν προβάλλεται αρκετά, δεν το γνωρίζει ο κόσμος, δεν ε, το ξέρουν αυτοί που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από το ταμείο αυτό και που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τις προπληρωμές που γίνονται από αυτό το ταμείο. Συχνά είναι τα μικρά προγράμματα, οι μικροί χρήστες εντό εισαγωγικών, που δεν μπορούν να χρημοδοτήσουν από τη δικιά τους ε, την πλευρά το κομμάτι το οποίο πρέπει να βάλουν για να μπορέσουν να πάρουν χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Προσπαθούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και αυτό θα ήταν σημαντικό. Θέλω ακόμα να υπογραμμίσω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην παρακολούθηση και στον έλεγχο. Βλέπετε συχνά οι λογαριασμοί, αποδείξεις, ελέγχονται και από τους ελέγχους αυτούς και τους υπολογισμούς διαπιστώνουμε τι μια φορά ότι τρία σαντίμ και έτσι η λογιστική διαδικασία ελέγχεται καλά, αλλά η ουσία μένει απ' έξω, δεν ελέγχεται το πραγματικό το ουσιώδες αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, να γίνεται ένας ουσιαστικός έλεγχος. Το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που εντοπίζονται έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά και με τα άλλα διορθωτικά ταμεία. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ρύθμιση του 50 διότι Δεν πρέπει να αναλύουμε σε βάθος το πρόβλημα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μετά να κάνουμε την ίδια περιγραφή και για άλλα ταμεία. Ζητάω λοιπόν κυρία Πρόεδρε από εσά να φροντίσετε να τηρηθεί το άρθρο 50 της διαδικασίας και με πιο ελαστικό τρόπο. Είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε καλές λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λέει Πρόεδρος. Θα δούμε τι δυσκολίες προκύπτουν δεν μου είχαν πει ότι υπήρχαν προβλήματα με την έκθεσή σας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η κυρία Χίρς τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Edith Bauer, την εισηγήτρια. Μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να έχει πολύ περισσότερη χρηματοδότηση, αλλά υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να εξάρω. Έχουμε συζητήσει και το θέμα σε μια σειρά από ομάδες εργασίες το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες χωρίς να επιβαρύνουμε την γραφειοκρατία. Πολλές φορές υπάρχουν μικρές ενώσεις, μικρές οργανώσεις ατόμων οι οποίες έχουν πολύ, πολύ λίγους πόρους και έχουν μεγάλο πρόβλημα να μπορέσουν να αποκομίσουν μια χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο λοιπόν και ίσως θα μπορούσε να υπάρξει μια προσθήκη σε αυτά που είπατε και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι ένα σημείο στο οποίο εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και επίσης να υπάρξει μια καλύτερη συγχρηματοδότηση από το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και χαίρομαι λοιπόν που μπορούμε και τώρα να δώσουμε ένα σαφές ε, μήνυμα στην Κομισιόν σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε το κοινωνικό ταμείο. Ο κύριος Τσαμπαωρή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η... Μερικές φορές υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία νομίζω ότι η γνωμοδότηση της κυρίας Μπάουερ τα ανατάμνει με τρόπο ιδιαίτερα ενδελεχή. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει όμως να μπορέσουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα προβλήματα. Εγώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε διατρέξει μακρόν δρόμο. Πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε τις διαβουλεύσεις σε σχέση με τη στρατηγική 2020 και τότε είχαμε την εντύπωση ότι όλη η πολιτική συνοχής θα έπρεπε να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Αλλά έκτοτε έγινε σαφές ότι έχουμε αρχίσει να εντοπίσουμε το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Και έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες από όλες τις πολιτικές παρατάξεις για να υπάρξει μια κοινή στάση και αυτές οι προσπάθειες απέφεραν καρπούς ο λίγων κατ' ο Είναι χρήσιμη λοιπόν πολύ αυτή η γνωμοδότηση και την εκτιμώ ιδιαίτερα. Χαίρομαι για την παράγραφο που αφορά το επίπεδο συγχρηματοδότησης, το ποσοστό συγχρηματοδότησης, γιατί όπως ελέγχθη είμαστε πολλές φορές ιδιαίτερα ε, λεπτομεριακοί και εξαντλητικοί για το αριθμητικό, για το για του αριθμού που περιέχονται στου λογαριασμού, χωρί να μα ενδιαφέρει η ουσία. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η υπερβολική αυστηρότητα και γραφειοκρατία η οποία αποτρέπει τελικά τους δυνητικού χρήστε. και αποδέκτες αυτών των κονδυλίων χρειάζεται και μια μεγαλύτερη ευκαμψία γιατί η κατάσταση μπορεί να ποικίλει κατά πολύ από τις πλούσιες περιοχές, τις περιοχές, τις φτωχές της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και υπάρχουν και περιοχές της Γαλλίας όπου υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα όπως την απόμακρη νήσο της Ρεουνιών. Τα πράγματα είναι διαφορετικά στην νήσο της Ρεουνιών από ότι στην νήσο της Γαλλίας, την Ile de France δηλαδή λέει ο μιλητής, κάνω ένα λόγο παίγνιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και συγχαίρω την Edit για την πολύ καλή αυτή γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε κύριε Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, είναι αλήθεια. Πολλά πράγματα έχω αφήσει απ' έξω στη γνωμοδότησή μου αυτή. Θα ήθελα να αναφερθώ στα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται συγχρόνως από πολλά ταμεία. Ε, δυστυχώς δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό. Παρόλο που είναι κάτι σημαντικό Πάντως, έχω εμπιστοσύνη στις συζητήσει που γίνονται στην ομάδα εργασίας. Ακούσαμε ότι το έγγραφο της Επιτροπής θα λάβει υπόψη και την πτυχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τους συναδέρφους για τις παρεμβάσεις τους. Περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τροπολογίες σας. Και εγώ θα υποβάλω τροπολογίες για τα θέματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ε, Όντω, τώρα που θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο τη διαδικασία, θα εμπλουτίσετε τη γνωμοδότησή σα αυτή με τροπολογίε. Οι τροπολογίε πρέπει να υποβληθούν πριν τι 3 Μαου στι 12 το μεσημέρι για να μπορέσουμε να τι εξετάσουμε στι 24 και 25 Μαου. 15 Ιουνίου θα εξετάσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες και 16 Ιουνίου θα ψηφίσουμε. Η Ρέγκη θα αποφανθεί και θα ψηφίσει δηλαδή στις 21 Ιουνίου. Δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Συνεπώς τελειώσαμε και θα τα ξαναπούμε στις 9 το πρωί στις 24 Μαΐου. Έληξε συνεδρίαση. Καλό βράδυ και ευχαριστώ πολύ όλους όσοι παρέμειναν μέχρι αυτή την ώρα στην αίθουσα. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει Πρόεδρος.